Uh, Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ήδη τρεις η ώρα. Uh, Οπότε, οι ελάχιστοι που είμαστε εδώ, ας εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Οι δύο δηλαδή. we'll have to wait because we've got Mr. Kansian and Mrs. Ayala Sender up, up first. Θα εξετάσουμε πρώτα την έκθεση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ. Yeah. Τώρα που έχουμε γίνει τέσσερις αγαπητοί συνάδελφοι, τουλάχιστον, κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης. Έχετε λάβει την ημέρη διάταξη. Την εγκρίναμε ήδη. Ε, συμφωνείτε? Ωραία. Τότε να πάμε στο δεύτερο σημείο, τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. Η συγκεκριτής είναι ο κύριος Αντώνιο αν Έχετε το λόγο. Grazie Presidente. Ehm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή την τελευταία περίοδο προσπαθήσαμε να συμφιλιώσουμε τις απόψεις με το Συμβούλιο. Αλλά αυτή η προσπάθεια είναι δύσκολη τελικά. Διότι η θέση του Συμβουλίου είναι αρκετά περιοριστική για αυτόν τον κανονισμό. Ξεκινούμε από την έγκριση σε πρώτη ανάγνωση. που βασίζεται σε ένα κείμενο του κ. Αλμπερτίνη, που είναι πολύ προστατευτικό, πολύ καλό για τους χρήστες. Η δουλειά λοιπόν που κάναμε και που προσπαθήσαμε να προωθήσουμε ήταν να μην υποχωρήσουμε και να μην αλλοιώσουμε την θέση που προέκυψε σε πρώτη ανάγνωση. Κατά διάρκεια αυτών των συζητήσεων και κατά διάρκεια αυτών των συναντήσεων προέκυψαν διάφορα επιχειρήματα για την αρχή της επικουρικότητας, για την συμμόρφωση με τον κανονισμό που εγκρίθηκε για τους ιδιοδρόμους και είδαμε το Συμβούλιο να έχει στάσει άκαμπτη, αμετακίνητη, ακλόνητη. Σε αυτή την δύσκολη οικονομική στιγμή λέει ότι δεν θέλει να υποσκάψει ας πούμε, την οικονομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα με τις επενδύσεις. Αλλά αυτό προσκούεται στην αρχή της ευθύνης των ιδίων των φορέων των μεταφορέων και την ε, δική μας την ε, αρχή, στα πλαίσια αυτού του κανονισμού, για τα δικαιώματα των χρηστών, των επιβατών. Το πρόβλημα προέκυψε στα... στο πεδίο εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Η συζήτηση για το πεδίο εφαρμογή αφορά τις παρεκκλήσεις που δίνονται στα κράτη-μέλη τα οποία μπορούν να μην λάβουν υπόψη τις περιφερειακές μεταφορές. Υπάρχει μια στεναρή θέληση του Συμβουλίου να αφήσει στα κράτη-μέλη αυτή τη δυνατότητα, παρεκκλήσεων δηλαδή. Εμείς λοιπόν, μαζί με την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιμείναμε ότι το πεδίο εφαρμογής δεν μπορεί να αφήνει εκτός του κανονισμού το 75% των μεταφορών με λεωφορεία. Η συμβαστική λύση λοιπόν θα μπορούσε να είναι να αφήσουμε εκτός τους περιφερειακούς μεταφορές και σε όλα τα μέσα μεταφοράς με λεωφορεία να συμπεριλάβουμε ένα πακέτο βασικών δικαιωμάτων που θα ισχύουν για όλες τις μεταφορές από τις αστικές μέχρι τις διεθνείς. Συζητάμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ποια είναι αυτά τα δικαιώματα, ποιο είναι αυτό το πακέτο, τι περιλαμβάνει αυτό το πακέτο, το οποίο θα πρέπει να ισχύσει για όλες τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν. Νομίζω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε μια συμβαστική πρόταση. Γιατί όλα μας τα επιχειρήματα για το πεδίο εφαρμογή βασίζεται και σχετίζεται με το άρθρο 2 παράγραφος 4. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιμείνουμε ότι πέρα από την, το να προασπίσουμε τα δικαιώματα των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα, ενημέρωση, κατάρτιση των υπαλλήλων και βοήθεια προς αυτούς τους ανθρώπους, να αποκλείσουμε από τις παρεκκλήσεις και τα δικαιώματα σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμών ή απώλεια των αποσκευών. Δηλαδή άμεση ευθύνη, άμεση ευθύνη που θα ισχύει χωρίς ο χρήστης, δηλαδή ο επιβάτης, να αναγκαστεί να προσφύγει σε οποιοδήποτε μηχανισμό ε, δικαστικό ή άλλο. Τώρα, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και ελπίζω ότι στις 6 του μηνός που θα γίνει ακόμα μια τριμερή συζήτηση θα καταφέρουμε να συμπληρώσουμε αυτά τα βασικά δικαιώματα, αυτόν τον κατάλογο με τα βασικά δικαιώματα που θα ισχύουν για όλους. Και εν συνεχεία, ξέρω ότι στις 6 Μαΐου στις 12 η ώρα είναι τελευταία ημερομηνία για τις ε, τροπολογίες και η ψηφίζει η Επιτροπή την 1η Ιουνίου και η Ολομέλεια την 1η Ιουλίου. Ελπίζω λοιπόν αυτά τα δεδομένα στις 6 του μηνός να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το συμβιβασμό. Γιατί ε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Παρά μόνο να εξασφαλίσουμε αυτά τα βασικά δικαιώματα. Δεν είναι αυτό που θέλαμε εμείς, μόνο τα βασικά δικαιώματα. Αλλά μόνο σε αυτό το ε, πεδίο, σε, αυτό το, σε αυτή τη βάση μπορούμε να καταφέρουμε να συμβαστούμε με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την προθεσμία για τις ε, τροπολογίες, Κάποιοι ευρωβουλευτέ ζήτησαν παράταση της προθεσμίας, γιατί παρά είναι βραχία. Γι' αυτό προτείνουμε να λήξει η προθεσμία σε 7 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Οπότε αν συμφωνείτε με την 7η Μαΐου κύριε Κάντσαν στις 12 το μεσημέρι ας παραταθεί λίγο η θεωρία για τις τροπολογίες ώστε να προλάβουν όσοι θέλουν να καταθέσουν τροπολογίες να το κάνουν. Όντως παρά είναι πολύ βραχή αυτή η προθεσμία γιατί στο μεταξύ είχαμε και διάφορες αργίες οπότε παραστένεψε το χρονικό περιθώριο. Γι' αυτό αν δεν έχετε αντίρρηση 7 Μαΐου 12 το μεσημέρι. Έχω πρόβλημα με τις 7 του μηνός Πρόεδρε. Έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να με δώσει 7 του μηνός. No, that would be the deadline for amendments. Perfetto. That would be for the deadline. Αυτό είναι για τις τροπολογίες μόνο. Ε, στις 7 λίγη διορία για τις τροπολογίες, όχι συζήτηση. Mrs. Meissner, sorry I forgot to put the mic on. Mrs. Meissner. Η κυρία Meissner. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο εισηγητής που έκανε, έκανε εδώ πέρα πολλή δουλειά, το γνωρίζω και τον ευχαριστώ και δεν ήταν απλό γιατί η πρόταση της ε, Κομισιόν και αυτά τα οποία είπε το Συμβούλιο ήταν τελείως διαφορετικά πράγματα. Και το ανέφερε ο κύριος Κάντσιαν πως ε, έχουμε τρίτο τριμερή διάλογο αυτή τη βδομάδα που ελπίζουμε να πετύχουμε κάποια πράγματα. Πράγματι είναι δύσκολο το θέμα εδώ σε δύο σημεία πρώτον το θέμα της συμπερίληψης ή μη των περιφερειακών μεταφορών με λεωφορεία που δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει. Το Συμβούλιο θέλει να εξαιρέσει τις περιφερειακές συγκοινωνίες, η Κομισιόν θέλει να τις συμπεριλάβει και εμείς έχουμε μια συμβαστική λύση που λέμε εκεί όπου υπάρχει ολοκληρωμένη υπηρεσία μεταξύ περιφερειακής και αστικής και προαστιακής κυκλοφορίας να συμπεριληφθεί. Αν δεν υπάρχει άμεση σύνδεση με αστική και προαστιακή συγκοινωνία να μπει στον κανονισμό, ενώ στην άλλη περίπτωση να εξαιρεθεί. Βέβαια αυτά τα πράγματα δεν είναι κάπως τόσο απλά σε όλα τα, τα κρατημέλη. Υπήρχε οι περιφερειακές συγκοινωνίες στη Γερμανία είναι αρμοδιότητα των κρατηδίων, οι πανεθνικές είναι αρμοδιότητα των σονδιακού κράτους, αλλά σημεία δεν γίνεται διάκριση, οπότε είναι θέμα των αρμοδιοτήτων εδώ πέρα να υπάρξει μια κοινή γραμμή, το ελπίζω. Τουλάχιστον και ένα άλλο σημείο είναι πράγματι αυτή η εξωτική πληρωμή, βεβαίως, εντάξει, να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των αναπήρων να έχουν πρόσβαση όπως και στο σιδηρόδρομο. Άλλωστε χρειάζονται και τις ανάλογες ε, πληροφορίες ε, με έναν αποδεκτό τρόπο αλλά βεβαίως πρέπει να δούμε και το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα πρακτικά, πώς θα εφαρμοστεί γιατί δεν είναι τόσο απλό στο λεωφορείο σε ένα λεωφορείο έτσι, περιφερειακής συγκοινωνίας ε, δεν μπορεί να ξέρει κανείς εκ των προτέρων εάν θα του έρθει ανάπηρος επιβάτης ή όχι. Αλλά πράγματι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση των αναπήρων και το θέμα μετά των αποζημιώσεων πηγαίνει πάρα πολύ μακριά στην πρόταση της ε, Κομισιόν. Πρέπει να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε λίγο τα πράγματα γιατί κατά την άποψή μου εδώ πέρα σωστά είπε το Συμβούλιο πως ε, σε αποζημιώσεις ε, πρέπει να δούμε και το εάν μπορούν να πληρώσουν τέτοια ποσά οι επιχειρήσεις. Π.χ. άτομα τα οποία είναι εξαρτημένα από κάποιον άλλο να συμπεριλαμβάνεται και αυτός εάν τραυματιστεί σε κάποιο ατύχημα διαβίου. Ναι, εντάξει, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των επιβατών, αλλά να διατηρηθεί και κάποια δυνατότητα, να μην απειλείται και η ίδια ύπαρξη των ε, εταιριών γιατί αντιλαμβάνομαι γιατί ε, προβάλλει αυτά τα επιχειρήματα το Συμβούλιο. Ελπίζω λοιπόν πέμπτη να βρούμε μια συμβαστική λύση και... Α, εγώ ζήτησα να παραταθεί και η προθεσμία των τροπολογιών γιατί αν έχουμε πρωί της πέμπτης ε, τον τριμερή διάλογο καλό είναι να μπορούμε και να αντιδράσουμε. Οπότε καλό είναι ε, μέχρι το μεσημέρι να μπορούμε να καταθέσουμε κάτι γραπτός, να παραταθεί λίγο δηλαδή η προθεσμία. Ευχαριστώ κυρία Λίχτεμπέργκερ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα κύριε Κάντσιεν, γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση με το Συμβουλίο, ειδικά όταν μιλάμε για εθνικές ιερές αγελάδες. Αλλά ένα πράγμα δεν αντιλαμβάνομαι. Είναι απέτηση και του κλάδου ειδικά όταν ε, αγοράζουν λεωφορεία να δουν και το πώς θα βοηθηθούν οι ανάπηροι. Αυτό ζητάει και ο κλάδος, να μην επιδοτείται δηλαδή μόνο η ιδιωτική αγορά γιόταχη για τους ανάπηρους. Οπότε εδώ πέρα δεν μπορώ να ακούω το Συμβούλιο να λέει πως όλα αυτά δεν γίνονται. Δεύτερον, όταν αποκλείουμε τις περιφερειακές συγκοινωνίες ε, και μετά έχουμε θεμελιώδη δικαιώματα που θα ισχύουν παντού. Το ερώτημα είναι πρώτον ποιος ελέγχει, δεύτερον υπάρχει προθεσμία και τρίτον ποιος έχει μετά την δυνατότητα να κάνει κάτι εάν δεν υπάρχει εφαρμογή. Υπενθυμίζω μόνο πως πολλά κράτη-μέλη έχουν την ελευθερία από ε, εμπόδια στην ομοθεσία τους και είναι επίσης συμβαλόμενα μέρη στην ομοθεσία για τους αναπήρους. Το έχει υπογράψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν όλα αυτά δεν είναι δεσμευτικά, απλά κάτι έτσι ωραίες δηλώσεις οι οποίες τελικά δεν εξυπηρετούν σε τίποτα, νομίζω πως... Ε, εδώ πέρα τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν κάποια κινητική δυσκολία ε, παραβιάζονται, περισσότερο τους βλάπτουμε. Οπότε θεωρώ πως πρέπει επιτέλους να τα πάρουμε σοβαρά αυτά τα πράγματα εάν ε, είναι να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή αυτό το πακέτο για μένα θα κριθεί από το κατά πόσον δεσμευτικό είναι. Υπάρχει κάποιος δηλαδή στα κράτη-μέλη που θα τους υποχρεώσει σε εφαρμογή ή είναι απλά ωραίες δηλώσεις ε, που είναι μόνο θεωρία και από πράξη μηδέν. Αυτός είναι ο φόβος μου εδώ πέρα. Έχουμε σε πάρα πολλά θέματα έλλειμμα εφαρμογής και θα έχουμε και το επόμενο που θα είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό φοβάμαι εγώ. Γι' αυτό ας είναι και μια δήλωση του Συμβουλίου που δεσμεύεται να αναπτύξει μηχανισμούς ελέγχου μεταξύ των κρατών μελών ή όπως αλλιώς θέλουν να το κάνουν. Αλλά μία δήλωση δικαιωμάτων που θα ισχύουν παντού τα έχουμε. Έχουμε συντάγματα, έχουμε συμβάσεις. Ε, τι γίνεται όμως. Έχουν γίνει ελάχιστα έως τίποτα όσον αφορά τα άτομα με κινητικές δυσκολίες για τα λεωφορεία. Τώρα όταν μιλάμε για τις αποζημιώσεις Καλό, εντάξει, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε ότι είναι μικρές επιχειρήσεις και δεν μπορούν να πληρώσουν, αλλά πρέπει να σα πω το εξή. Εάν αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει το δικαίωμα μόνο και μόνο γιατί είναι μικρή η επιχείρηση, τότε θα χάσουν και αυτοί οι άνθρωποι και οι μικρές επιχειρήσει. επιχειρήσεις και βέβαια οι πολίτες που δεν θα έχουν ε, πλέον αυτά τα δικαιώματα. Τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω Βεβαίως εδώ πέρα έχουμε την ε, τη μία υπηρεσία εδώ πέρα που θα φροντίσει για την ε, εφαρμογή και δεν αναφέρεται πως είναι ανεξάρτητη. Ελπίζω να είναι ανεξάρτητη γιατί αυτό για εμένα βεβαίως είναι ξεκάθαρο. Εάν αυτή η υπηρεσία δεν είναι ανεξάρτητη, εάν καταφεύγει κανείς εκεί, κάνει παράπονα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα και τον στέλνουν ε, από τον Άννα στον Καϊάφα, ε, θα είναι τελείως αρνητική η κατάσταση και θα επηρεάσει τελείως αρνητικά τα δικαιώματα των επιβατών. Αυτά για μένα είναι σημεία χωρίς επιστροφή και από αυτά θα εξαρτηθεί η συμφωνία μου. Δηλαδή, ε, επίσης, όταν εάν δεν θέλουν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτή την νομοθεσία, εάν τα αναβάλουν, εάν ισχύσει μόνο για κάνα δύο λεωφορεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, τότε θα έχουμε εσπαταλήσει και το χρόνο μας για να μην γίνει τίποτα στο τέλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να υποστηρίξω αμέριστα τις βασικές αρχές των μέτρων που προτείνονται. Αλλά όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και όπως είδαμε και με άλλους κανονισμούς για, τα, για τις αποζημιώσεις, η αρχική πρόταση ήταν μια οριζόντια πρόταση από το σιδηροδρομικό πακέτο και τώρα επεκτάθηκαν οι αποζημιώσει ε, και στις οδικές μεταφορές και στις θαλάσσιες. Θα πρέπει να γίνει όμω διάκριση μεταξύ των διαφόρων, γιατί δεν πρέπει να τα βάζουμε όλα στην ίδια σκάφη. Για παράδειγμα, οι αποζημιώσει για τις αεροπορικές, τις ιδεοδρομικέ μεταφορές και τα δικαιώματα που κατοχυρώνται για του επιβάτε είχαν συγκεκριμένη μορφή αλλά δεν είναι το ίδιο για τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν, ιδιαίτερα για τις ε, αστικές ή προαστιακές. Γιατί ακόμη και ανακυρωθεί ένα δρομολόγιο, μετά από 10 ακολουθεί άλλο. Δεν ξέρω, ίσως για τι αγροτικέ ε, περιοχές, αγροτικές όχι τόσο, αλλά δεν είναι το ίδιο αυτό που ισχύει στις οδικές μεταφορέ, με λεωφορεία και πούλμαν από ότι στι αεροπορικέ, για παράδειγμα ή στις σιδηροδρομικέ. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε και από τις δύο προλαλήσασες είναι το θέμα της ευθύνης σε ασφαλιστικές εταιρείες και τα πακέτα αποζημιώσεων. Γιατί για τις μικρές επιχειρήσεις δεν θέλουμε να τις καταβαραθρώσουμε. Γιατί πολλές μικρές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν τέτοιες προαστιακές ή περιφερειακές συγκοινωνίες. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ειδικέ ρυθμίσει για τέτοια επίπεδα αποζημιώσεων και να είμαστε πρώτα απ' όλα ρεαλιστέ και πρακτικοί. Εγώ είμαι υπέρ της θέσης του Συμβουλίου. Και δεν νομίζω ότι είμαι θεροβάμων, γιατί ιδιαίτερα σε αυτό που είπαμε για τις ε, αστικές και προαστιακές συγκοινωνίες, προτιμώ να περιορίζονται ρυθμίσεις ε, στις ε, διεθνείς μεταφορές, διασυνοριακές. Γιατί αν αρχίσουμε να ρυθμίζουμε τα πάντα μέχρι και τις τοπικές ε, υπηρεσίες μεταφορών με λεωφορεία, θα δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσουμε. Και όπως είπε η κυρία Λίχτεμπεργκ, θα είναι και ανεφάρμοστα ένα τέτοιο μέτρο. Μπορεί να είμαι κάπως απομονωμένο στη θέση αυτή, αλλά ελπίζω αυτή τη φορά να συμφωνήσουμε ότι τουλάχιστον περιορίζεται μόνο στις διεθνείς μεταφορές, στα διεθνή δρομολόγια. Okay, thank you, thank you. Mr. Κύριε ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Η Ντέμπορα Σερατσίνη, η σχεδοσυγήτρια, δεν μπόρεσε να έρθει, οπότε στη θέση της θα ευχαριστήσω εγώ τον εισηγητή για την καλή συνεργασία Υπάρχουν κάποιες ε, παρατηρήσεις που συμφωνούν ε, με αυτά τα οποία ήδη ακούστηκαν όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής ε, νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε πράγματι στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων οπότε οι αστικές μεταφορές να μείνουν εκτές επίσης πρέπει να έχουμε ένα καλό ορισμό βεβαίως για το τι σημαίνει περιφερειακές ειδικά μεταφορές όταν μιλάμε για τις μεγάλες αποστάσεις γιατί πρέπει να φύγει εδώ πέρα αυτή η ασάφεια. Υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες ε, στην ερμηνεία τώρα καταγγελίες ε, και αποκατάσταση. Πράγματι το βάρος αποδείξεως πρέπει να είναι ε, στον επιβάτη. Πρέπει να δούμε βέβαια και τα πράγματα από τη μεριά του γιατί πιθανότητα αυτό είναι το θύμα. Επίσης διαπιστώνει η σκιώδη συγγήτρια πως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τις επιδοτήσεις γιατί υπάρχει η δυνατότητα απάτης. Να δούμε δηλαδή τι έχουμε κάνει με τα δικαιώματα των επιβατών τρένων και να βρούμε μια ανάλογη ρύθμιση γιατί είναι ανάλογη και η κατάσταση. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για την ομάδα μας είναι βεβαίως ε, αφορά τους ανθρώπους ε, που έχουν, ε, είναι εξαρτημένοι από κάποιους άλλους και να υπάρχει βεβαίως η ανάγκη συμπαράστασης, να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα 20 24 ώρες βοήθειες Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό για ένα ταξίδι με λεωφορείο και επίσης σημαντικό είναι να δούμε την απομάκρυνση εμποδίων στην υποδομή, σταθμού των λεωφορείων, όπως ακριβώς γίνεται και για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Αυτά. Κατά λοιπά, σε γενικές γραμμές νομίζω είμαστε στην ίδια γραμμή. Ευχαριστώ κύριε Γκρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτά τα οποία έχει κάνει μέχρι στιγμής. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση εδώ πέρα γιατί όλοι είναι υπέρ των δικαιωμάτων των επιβατών και ειδικά αυτών με μειωμένη κινητικότητα. Από την άλλη βεβαίως προσπαθούμε να συμβάσουμε την αρχή της αναλογικότητας εδώ πέρα και μιας λογικής ε, εφαρμογής των πραγμάτων. Γιατί αυτό το οποίο θέλουμε τελικά είναι το συμφέρον των επιβατών και όχι των δικηγόρων. Οπότε προβλέματα τα οποία αναγνωρίζουμε ήδη πρέπει ήδη τώρα στη ρίζα να αντιμετωπιστούν. Όσον αφορά λοιπόν το πεδίο εφαρμογής ε, δεν ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μικρό γιατί αφενός δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρό γιατί θα είναι ανεφάρμοστο και γιατί σε μικρότερες περιοχές επίσης συχνά υπάρχει μια κινητικότητα με πάρα πολλά μέσα και θα οδηγηθούμε στην εξής ε, παράλογη κατάσταση. Εάν υπάρχει άμεση σύνδεση διαφορετικών μέσων μεταφορών μπορούμε να οδηγηθούμε σε καθυστερήσεις που αυτομάτως οδηγούν σε αποζημιώσεις κτλ. Να το δούμε δηλαδή ρεαλιστικά, όχι μόνο στην θεωρία. Να επιθυμίσω τώρα για τους συναδέλφους που μιλάνε για μεθοριακές περιοχές. Υπάρχουν αποστάσεις 10 χιλιόμετρων που καλύπτονται από δύο συνοριακές γραμμές ακόμα και με μετρό, με υπόγεια δίκτυα έχουμε δύο συνοριακές γραμμές. Οπότε πρέπει να το δούμε τι γίνεται επί τόπου. Δηλαδή το να λέμε διεθνείς μεταφορές δεν σημαίνει ότι είναι πάντα τόσο μεγάλες οι αποστάσεις ε, ε, ε. όσον αφορά τώρα τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή πώς πρέπει να γίνουν οι διάφορες ε, διαδρομές βεβαίως προσβάσιμα για τα άτομα αυτό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στο κάθε όχημα ε, υπάρχει όντως αυτή η ανάγκη και η ζήτηση. Δηλαδή δεν το βρίσκω σωστό να υπάρχει μια γραμμή που δεν θα είναι ε, προσβάσιμη, αλλά δεν το θεωρώ σωστό να είναι και κάθε όχημα σε κάθε γραμμή, ειδικά μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις ε, να έχει αυτή την υποδομή, αν δεν υπάρχει τακτική ζήτηση. Δεν ξέρω, θα μπορούσε να δημιουργηθεί εδώ πέρα ένα αποδεματικό. Ελπίζω πως θα πρέπει να το δούμε αυτό λογικά και να δούμε και το τι σημαίνει επιτόπου ή αν είναι εφικτές αυτές οι λύσεις ή όχι και να λάβουμε υπόψη τις μικρές επιχειρήσεις. Μία μικρή επιχείρηση με ένα-δύο άτομα δεν μπορεί να εγγυηθεί την φυσική συνοδεία κάποιου ε, σε ένα μεγάλο αριθμό λεωφορείων. Αν είναι δηλαδή να εξαφανίσουμε τις μικρές επιχειρήσεις, να το πούμε. Και εδώ πέρα μπορούν, εγώ θεωρώ, να υπάρξουν μικρές επιχειρήσεις και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των επιβατών, εάν βρούμε μια καλή λύση. Ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνικός. Καταρχήν, όπως είπε ο κύριος Γκρό, θα πρέπει να μην είμαστε υπερβολικά σχολαστικοί και να στοχεύσουμε τις μικρές επιχειρήσεις. Ούτε ως προς τα δρομολόγια, ούτε ως προς το, τη διαστάσεις. Και όταν λέμε περιφερειακές, άλλο περιφερειακές μεταφορές με λεωφορείο και άλλο περιφερειακές με αεροπλάνο. Πώς θα το ορίσουμε το περιφερειακές συγκοινωνίε, Γιατί μερικοί δεν θέλουν να, να καλύπτονται οι περιφερειακές μεταφορές ε, και να κατοχυρώνονται και τα δικαιώματα των επιβατών, ενώ μερικέ φορέ οι περιφερειακές είναι σαν προαστιακές. Θα πρέπει να δούμε πού θα βάλουμε τη διαχωριστική γραμμή. Κάτι που είχα πει και στην προηγούμενη μα συνεδρίαση και στην προηγούμενη επιτροπή, αν μπορούμε να έχουμε έναν νέο χάρτη των δικαιωμάτων των επιβατών στην Ευρώπη, θα είναι και πιο κατανοητός για τους πολίτες, πιο εύληπτος, ε, γιατί τα έχουν χάσει λίγο με τόσες πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις που ισχύουν για κάθε μέσο μεταφοράς. Και θα μας βοηθήσει ένας τέτοιος ενιαίος χάρτης, μια τέτοια ενιαία χάρτα. Μπορούμε να έχουμε ξεχωριστά πρωτόκολλα, αλλά τουλάχιστον μία δέσμη κανόνων να είναι κοινή και θα μας βοηθήσει και το είπε και ο Αντώνη ότι και εκείνο ήταν πιο σαφή στο έργο του. Θα μπορούσαμε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, επανεξετάσουμε το θέμα τη... του κοινού σώματος διατάξεων ε, για τα δικαιώματα των επιβατών με επιμέρους πρωτόκολλα για τα διάφορα είδη μεταφοράς ίσως. Ο κύριος Κόζακ Köszönöm a szót. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőknek. Να ευχαριστήσω του συζητητές για αυτή τη στεναρή θέση που μας παρουσίασαν και για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των επιβατών. Θα ήθελα να κοιτάξω αυτό το θέμα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Όταν μιλάμε για άτομα με αναπηρίες, με ειδικέ ανάγκες, Ίσως αυτός ο ορισμός δεν καλύπτει και άλλες περιπτώσεις, όπως ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή ε, ανθρώπους με πολύ μικρά παιδιά ε, ή ανθρώπους που έχουν ε, ακουστικά προβλήματα ή ξένους που δεν γνωρίζουν την τοπική γλώσσα. Όταν μιλάμε λοιπόν για ανθρώπους με αναπηρίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, για τα 50 εκατομμύρια Ευρωπαίων που έχουν αναπηρία στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες. Γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω στους ε, εισηγητές τουλάχιστον η τροπολογία 11, 12, 13 και 14, 22, 23 και 35, αυτές οι τροπολογίες να γίνουν τουλάχιστον αυτές αποδεκτές, το ελάχιστο είναι να προσφέρουμε κάποια δικαιώματα ε, στους ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες, με αναπηρίες. Υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Ο ρόλος του κράτους το κράτος, η κυβέρνηση πρέπει να παίξει και, αυτή, και αυτό το ρόλο του. Και θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείε που εξασφαλίζουν τις μεταφορές βοηθούνται ούτως ώστε να είναι προσπελάσιμες, προσπελάσιμα τα μέσα μεταφοράς. Θα πρέπει λοιπόν στο κείμενο να πούμε ότι το κράτος πρέπει να παίξει ένα ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί αυτό το βάρο αυτό δεν θα πρέπει να το φέρουν μόνο οι εταιρείε. Θα πρέπει να το μοιράσουμε αυτό το βάρο και θα πρέπει και η κυβέρνηση να παίξει και αυτό το ρόλο τη να αναλάβει και αυτή αυτό που οφείλει να αναλάβει. Κοιτάξτε, εγώ απορώ πάντα που είναι τόσο δύσκολα αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη. Εγώ σας είχα πει, όπως είπα, σε κάθε λεωφορείο που είτε ταξιδεύει 2 είτε 5 είτε 100 χιλιόμετρα ε, είναι διάταξη να έχει πρόβλεψη για ανάπηρους. Γιατί? Λόγω των πολλών αναπήρων που υπήρχαν από το Βιετνάμ και τα λοιπά που δεν έπρεπε να αποκλειστούν. Εντάξει, εμείς μπορούμε να έχουμε τόσους πολλούς ανάπηρους πολέμου. Ε, δόξα τω Θεώ δεν είχαμε τόσους πολλούς πολέμους αλλά έχουμε ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα και αν μπορούν οι Ηνωμένε Πολιτείε να πούνε πως εμείς αυτό θα το, θα το επομιστούμε γιατί 30% των επιβατών εκεί πέρα είναι άτομα με κινητικές δυσκολίε. Ε, μπορεί να είναι ξέρω κάποιος στο πόδι του στο, κάνοντας σπορ είναι φοβερή εμπειρία υπάρχουν επίσης ε, καθηγητές ε, στη Βιέννη που διδάσκουν στους αναγκάζουν τους φοιτητές συγκοινωνιολογίας εκεί πέρα να περνάνε 15 μέρες σε μια αναπηρική καρέκλα για να δούνε πώς είναι. Και να λέμε πως αυτό πρέπει να γίνει μόνο στα μεγάλα ταξίδια γιατί αλλιώς δεν αξίζει ο τόπος. Όχι, πρέπει να είναι μια αρχή για να δείξουμε και την αλληλεγγύη μας με αυτούς τους ανθρώπους ε, και να τους λαμβάνουμε υπόψη γιατί ο καθένας θα μπορούσε να είναι. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι τώρα γιατί το τυραννάμε τόση ώρα. Υπάρχει και στις αεροπορικές συγκοινωνίες μόνο ευθυνές εταιρείε να κατά και λέγανε κόστος κτλ. Όχι, είναι αλληλεγγύη Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι και τα επιχειρήματα για αυτά τα οποία λέτε. Δηλαδή αυτό το οποίο μπορεί να κάνουν και είπα, εν πάση μπορεί να είναι αδύνατο στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Γέγκερ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά λακωνική. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κάντσιαν, τον εισηγητή, για τις ε, άοκνες προσπάθειες του και την σύστασή του που μας βρίσκει σύμφωνος και ως προς το πεδίο και ως προς την ευθύνη. Και συμφωνούμε ότι το καλύτερο είναι η χρυσή τομή. Εκεί θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία, μια συμβαστική λύση δηλαδή και ευελπιστούμε ότι στις 6 θα είναι ικανοποιητική η συμβαστική λύση, κυρίως ε, θα αποβαίνει προς όφελος των επιβατών. Θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένα σημεία που αναφέρθηκαν. Κύριε Μπράντμπερν, δεν προβλέπεται αποζημίωση στην πρόταση αυτή. Ούτε καμία προκαταβολή, κύριε Αλκαντράουι, δεν προβλέπεται. Και μάλιστα από τη στιγμή που το άρθρο 27 θα περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού 424, γιατί αυτό επισημάνεται ως ανησυχία, θα διασκεδαστεί αυτή η ανησυχία σας για τους ελέγχους, γιατί θα υπάρχει ανεξάρτητος φορέας και θα κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία του στον κανονισμό. Τεράστια ήταν η πρόοδος που συντελέστηκε και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να πω ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες να διευκολύνουμε την επίτευξη λύσης και να βρούμε μια ικανοποιητική συμβαστική λύση στη δεύτερη ανάγνωση. Τέλος, όπως δήλωσε ήδη ο Αρμόδιος Επίτροπος, συμφωνεί ότι ίσως ε, έχει οριμάσει η κατάσταση για τη χάρτα των επιβατών, αλλά σε ολοκληρώσουμε πρώτα το έργο μας για τις διάφορες μεταφορές, να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα για τις οδικές μεταφορές, μελοφορία, πούλμαν και μετά για τις ε, θαλάσσιες και μετά θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα για όλα τα μέσα μεταφοράς στον ενιαίο χάρτη. Ο εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν. Τους ευχαριστώ για τις συνεισφορές τους στη σημερινή συζήτηση. Και θα λάβω υπόψη όλα όσα άκουσα. Αυτό που θέλω να τονίσω, Πρόεδρε, είναι ότι προχωρούμε ε, προσπαθώντας να βρούμε τη σωστή συμβιβαστική λύση ανάμεσα στην ευθύνη των μεταφορικών εταιριών, γιατί δεν πρέπει να μπλέκουμε την έννοια της ευθύνης, με άλλου τύπου ευθύνες που θα μπορούσαν όντως να δημιουργήσουν ε, οικονομικά προβλήματα, ειδικά στις μικρομεσαίες ε, εταιρείε. Να βρούμε λοιπόν αυτή τη σωστή συμβιβαστική λύση, να του πούμε πρέπει να αναλάβετε περισσότερες ευθύνες, αλλά χωρίς να σας επιβαρύνουμε περιτά. Αυτή την ισορροπία προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε σήμερα για να τηλεσφορήσει αυτός ο κανονισμός. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ξεκινάμε από ένα κανονισμό ο οποίος εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση με έτσι πολύ έντονο και στεναρό τρόπο από εμά και από την άλλη υπάρχει ε, το αντίβαρο που είναι το Συμβούλιο που έχει και το ίδιο την ε, δική του έτσι έντονη θέση και προσπαθεί να υποσκάψει τη δική μας. Τώρα, ο στόχος μας ποιος είναι. Τι θα κάνουμε, θα κολλήσουμε στον όρο ε, περιφερειακός ή θα προτείνουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δηλαδή να προωθήσουμε ένα πακέτο από βασικά δικαιώματα που περιλαμβάνουν όλα όσα είπαν οι διάφοροι βουλευτές. Δηλαδή, περιλαμβάνουν και τους ανθρώπους ε, με κινητικά προβλήματα, ακόμη και αν έχουν προσωρινά κινητικά προβλήματα. Γνωρίζοντας ότι τους σταθμούς και τα λεωφορεία ε, που υπάρχουν ήδη δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, δεν μπορούμε να τα επηρεάσουμε γιατί αυτό ξεπερνά, υπερβαίνει τις, ε, την αρμοδιότητά μας. Επίσης υπάρχει και το θέμα του ενιαίου εισιτηρίου, one ticket, που το βάλαμε σε ένα εκτιμώντας. Αυτά για τα, για τα νέα μέσα να, να σεβαστούν δηλαδή τις ε, κοινοτικές διατάξεις που πρόκειται να προκύψουν. Αλλά μιλάμε τώρα για νέους σταθμούς, για νέα, νέες μεταφορικές εταιρείες, ε, όχι για τις ισχύουσες. Σε αυτή τη φάση λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου ενημερώνεται ο επιβάτης ε, υποβοηθείτε όταν το χρειάζεται και σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο έχει αυτές, αυτά τα δικαιώματα. Εν συνεχεία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω σε σχέση με τις διαπεριφερειακές και διασυνοριακές μεταφορές, ε, αφήνοντας στην άκρη το, τον όρο περιφερειακός. Η Κομισιόν αναφέρθηκε στο άρθρο 27 του κανονισμού και παρέπεψε σε αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να παραπέμψουμε και στον 2006 κάθος 2004, που αναφέρεται και στα εκτιμώντας. Παραπέμποντας λοιπόν και σε αυτόν τον κανονισμό, θα καταφέρουμε τελικά να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Αν καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε και τις περιφερειακές μεταφορές ε, συνδέοντάς τις με τις αστικές και προαστιακές. Το βασικό είναι να εξασφαλίσουμε αυτό το πακέτο δικαιωμάτων. Αν δηλαδή είναι ε, να θυσιάσουμε το, το... το θέμα των περιφερειακών μεταφορών για να εξασφαλίσουμε το βασικό πακέτο, το κάνουμε. Ευχαριστώ όλους όσους ε, συμμετείχαν. Την κυρία Λίχτεμπεργκ, την κυρία Μάισνερ, την κυρία Σερακιάνη, που ήρθαν μαζί μου για να συζητήσουμε αυτόν τον κονισμό. Κάτι που φαινόταν εκ πρώτη όψεως απλό, αλλά απεδείχθη ότι δεν ήταν τόσο απλό. Μετά από όλα όσα έχουμε πετύχει για τα άλλα μεταφορικά μέσα και σε σχέση με αυτά που θα ακούσουμε σε, σε λίγο από τη συνάδελφο που ασχολείται με τις θαλάσσιες α, μεταφορές, α, νομίζω ότι μπορούμε μετά από όλα αυτά και όσα πετύχουμε για το δικό μας θέμα για τα λεωφορεία και τα πούνα, μπορούμε να περάσουμε στο θέμα αυτού του, του βασικού χάρτη. Μεσημέρι 7 Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες. Είναι Παρασκευή. Θα ψηφίσουμε, ελπίζω, τον Ιούνιο και στην Ολομέλεια στην, τον Ιούλιο, 10 Ιουλίου. Πάμε τώρα στα δικαιώματα επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές με την κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και ο συνάδελφος Καντζάν, και στη δική μου περίπτωση έχουμε μια νέα κατάσταση. Στην πρώτη ανάγνωση χρειάστηκε να χειριστούμε την πρόταση του Συμβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την κυρία Βόρτμαν Κόλ, την κυρία Βόιλ, Λίχτεμπεργκερ, τις κοιόδης ηγήτριες ε, που μου συμπεραστάθηκαν προκειμένου να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις πρώτες συνομιλίες με την Ισπανική Προεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά το Μάθιο από τη Γραμματεία για την διευκόλυνση που μας έκανε και τη συνδρομή που μας παρήχε και να ευχαριστήσω και την Επιτροπή για τις προτάσεις της, παρόλο που μερικές φορές δεν μας διευκόλυνε όσο χρειαζόμασταν. Αλλά είχαμε κάποιους περιορισμούς στα δεδομένα, γιατί χρειαστήκαμε στοιχεία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών. Και ευχαριστώ και την Ισπανική Προεδρία που και αυτή έκανε ό,τι μπορούσε για να μπορέσει να παρουσιάσει καλύτερα τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους συναδέλφους του Συμβούλιο και να την κάνει αποδεκτή. Ο νευτιλιακές μεταφορές ε, έχει προχωρήσει, ο των ναυτιλιακών μεταφορών έχει προχωρήσει πολύ, ιδιαίτερα με τις κρουαζιέρες, γιατί πολλοί επιβάτες και τουρίστες χρειάζονταν αυτή τη σύγκληση και τις προσαρμογές αυτές. Υπάρχει μεγάλη πρόοδο στον τομέα αυτό των θαλάσσιων μεταφορών, αλλά θα πρέπει να προβλέψουμε ένα ομοιόμορφο πλαίσιο, ώστε για όλο τον κλάδο να υπάρχει εγγύηση και προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών. Υπήρξε αρκετή σύγκληση μεταξύ των θέσεων του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το λέω αυτό με ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί υπήρξε και προσέγγιση και ένα μεγάλο τμήμα των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναγνωρίστηκαν τουλάχιστον από το Συμβούλιο και έγινε μια προσπάθεια ε, ενσωμάτωσης του στο κείμενο, ακόμη και για θέματα που αρχικά υπήρξε μεγάλη διάσταση απόψεων. Παρόλα αυτά, απομένουν ε, σημαντικές διαφορές, εκκρεμούν πολλά σημεία, αλλά συνεχίζεται ο διάλογος για να συνεχίσουμε την προσέγγιση με το Συμβούλιο. Το θέμα του πεδίου εφαρμογή είναι από τα πιο επίμαχα, γιατί εκεί το Συμβούλιο φυσικά επηρεάζεται από τις τεράστιες διαφορές που υπάρχει στον τομέα αυτό στα 27 κρατη Γι' αυτό και μας πρότεινε ένα πεδίο εφαρμογή πολύ πιο περιορισμένο από αυτό που επιθυμούσαμε εμείς, αποκλείοντας όλα τα πλοία που είναι... που έχουν χωρητικότητα, χωρητικότητα μικρότερη από 36 επιβάτες. Εμείς ζητούσαμε 12 επιβάτες όριο, το Συμβούλιο 36. Επίσης, ε, ε, αποκλείστηκε από το Συμβούλιο τα πλοία με πλήρωμα λιγότερο από, τρι, από τρεις ανθρώπους ή ε, τα πλοία λιγότερα από 15 μέτρα ή και κάποια σκάφη αναψυχής, όχι τα καιρός γερόπλια, που σε μερικές περιπτώσεις εξυπηρετούν μεταφορές στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Γιατί και οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές διανύουν μια πολύ σημαντική κρίση δυστυχώς και από αυτή την άποψη η κοινή θέση προστατεύει τον κλάδο και εγώ θα συνεχίσω να υπερασπίζω τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο. Τώρα για, το, για τη διαφορά μεταξύ 12 και 36 επιβατών, εκεί υπάρχει μεγάλο περιθώριο. Θα προσπαθήσουμε να συγκλίνουμε κάπως τα πράγματα. Επίσης, το Συμβούλιο πρότεινε επιπλέον εξαίρεση για πλοία λιγότερο από 300 τόνους χωρητικότητα. Και η εξαίρεση αυτή δημιουργεί τεράστιες περιπλοκές και αβεβαιότητα, γιατί θα πάει ο κάθε επιβάτης να ρωτήσει αν η χωρητικότητα του πλοίου είναι πάνω από 300 τόνους και πώς έχει καταχωρηθεί. Λίγο δύσκολο το βλέπω πιστεύω ότι ακόμη και εκεί θα μπορούσαμε να διαβρύνουμε κάπως το πεδίο εφαρμογής. Μία σημαντική τροποποίηση που έγινε είναι τα άρθρα για τη συνδρομή, την αποζημίωση και την αποκατάσταση. Εκεί με κάποιες μικροπροσαρμογές είμαι βέβαια ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Υπάρχουν ε, αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν ως προς προθεσμίες, ε, ως προς τις ε, του ανθρώπου με κάποιε ειδικέ αναπηρίες ή προβλήματα κινητικότητας. Αυτό που μα χωρίζει με το Συμβούλιο είναι το θέμα του κατοφλίου κάτω από το οποίο δεν καταβάλλεται ουδεμία αποζημίωση. Εκεί το Συμβούλιο γνωρίζοντα την πυχμή και την αιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό έφτασε στο ανώτατο όριο των 40 ευρώ που, καλύπτει τους, που αποκλείει τους άλλους τα περισσότερα δρομολόγια. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε σε 16 ευρώ το μέγιστο κατόφλι, όπως έγινε και στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Επαναλαμβάνω το Συμβούλιο, επειδή ακριβώ αντιμετώπισε τις διαφορετικές καταστάσεις, χρειάστηκε να περιλάβει το θέμα των λιμένων, γιατί υπάρχουν τεράστια διαφορές μεταξύ των λιμένων και των υπηρεσιών που προσφέρουν. Οπότε από αυτήν την άποψη το επίπεδο προσφοράς υπηρεσιών των επιβατών είναι πολύ διαφορετικό. Από αυτή την άποψη πάντως ε, προχωρήσαμε με το Συμβούλιο και μάλιστα το ξεπεράσαμε ε, λάβαντος υπόψη και την έννοια του τερματικού λιμενικού σταθμού. Πάντως συνεχίζονται οι συζητήσεις με το Συμβούλιο. Επίσης προτάθηκε και το θέμα των 100.000 μετακινήσεων επιβατών για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος προκειμένου να προβλεφθούν ε, κάποιες προδιαγραφές ποιότητας. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει το κατόφλι να είναι οικουμενικό, δηλαδή και κάτω από 100.000 μετακινήσεις επιβατών ε, εφαρμόζονται αυτές οι προδιαγραφές ποιότητας. Αλλά πιστεύω ότι σε τέτοιου είδου μικροδιαφορές θα υπάρξει σύγκληση με το Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίε μου, που έχουν πια μεταφραστεί, επιχειρούν ε, να κρατήσουν ανοιχτό το διάλογο με το Συμβούλιο, ζητώντας όμως ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογή. Εγώ εμιένω στο αρχικό όριο της Επιτροπής των 12 επιβατών, παρόλο που σε ορισμένε περιπτώσεις ε, περιορίσαμε τις απαιτήσει μας. Για παράδειγμα, 4 ευρώ για το ελάχιστο κατόφυλλο. αποζημίωση και θα γίνει κάποια ελπίζω προσέγγιση με το Συμβούλιο. Επίσης το θέμα του βάρους απόδειξης ό,τι αφορά τις συνθήκες για τις οποίες ε, ε, αρνείται κάποιος την επιβίβαση, το βάρος απόδειξης θα το φέρει ο μεταφορέας. Όπω συμβαίνει και στι ενέργειε μεταφορέ. Γιατί εκεί είναι εύκολο ο πύργο ελέγχου να αποφασίζει. Αλλά στην περίπτωση των λιμενικών μεταφορών αποφασίζει ο καπετάνιο. Και ίσω ε, σε ορισμένε περιπτώσει υφίσταται τι πιέσει των εταιριών μεταφορά. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει σε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησης επιβίβασης το βάρος απόδειξης να το φέρει ο μεταφορέας. Για το σύστημα των παραπώνων και καταγγελιών. Εκεί ήταν θετική η θέση του Συμβουλίου να είναι ανεξάρτητος οργανισμός, να ισχύει ένα διπλό σύστημα, ώστε τα κράτη που έχουν δύο επίπεδα παραπώνων και καταγγελιών να παραμένουν αλλά ο οργανισμός αυτός να είναι ανεξάρτητος και η ανεξαρτησία του κατοχυρώθηκε στο κανονισμό. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών με περιορισμένη κινητικότητα ή αναπηρίες, εγώ με τις τροπολογίες μου ε, μίλησα για τα προσβάσιμε τις προσβάσιμες μορφές και τρόπους μεταφοράς, τις υποχρεώσεις, τις προθεσμίες, γιατί και εκεί υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο εργάσιμων ημερών που απαιτεί το Συμβούλιο και τις 48 ώρες που ζητούμε εμείς. Γιατί είναι πιο λογικέ 48 ώρε. Οι δύο εργάσιμε μέρε θα μπορούσαν να γίνουν 4 μέρε, αν μεσολαβήσει Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα. Γι' αυτό και προτιμώ τι 48 ώρε. σε περίπτωση των προθεσμιών καταγγελιών και εκεί περιορίσαμε, συντμήσαμε τι προθεσμίε γιατί από τη στιγμή που έχει περάσει ένα, μια μισή ώρα επιβάτης περιμένοντας τον τερματικό λιμενικό σταθμό, λογικό είναι να χρήζει κάποιες ε, συνδρομής, ανάλογα με το είδος των επιβατών που καταφθάνουν εκεί. Διατήρησε την τροπολογία 48. Περιλαμβάνεται αυτό το θέμα της διοικητικής αρρωγής του σημείου 40, στην τροπολογία 42 Επίσης προσθέσαμε και τα θέματα υγείας ό,τι αφορά την ασφάλεια για την άρνηση επιβίβασης. Βέβαια στις συζητήσεις που είχαμε από τους, με τους σκιώδεις ηγητές μέχρι στιγμής δεν επίστηκα για την ανάγκη προσθήκης και των λόγων υγείας πλέον τον επιπλέον στους λόγους ασφάλειας. Γιατί αν προσθέσουμε και την υγεία ως λόγο άρνησης θα ανοίξουμε ένα κουτί της πανδώρας. γιατί αν ζητούμε ιδιαίτερα συμπλήρωση περισσότερων διατυπώσεων ε, για θέματα υγείας, νομίζω ότι ανοίγουμε πραγματικά τους οσκούς του αιώλου, κάτι που είναι πρωτοφανές και δεν επιβλήθηκε σε κανένα τρόπο μεταφοράς. Γιατί να το προσθέσουμε στις πλωτές μεταφορές της θαλάσσιας. Από τη στιγμή που θα καλύψουμε και τους ε, τέσσερις τομείς ξεχωριστά, θα μπορούσαμε ίσως να καταλήξουμε σε μια πιο ε, συνεκτική ρύθμιση και δέσμη μέτρων κάτι που συνάδηκε με την επιθυμία μας για τη διαλειτουργικότητα, αλλά αυτό θα γίνει αργότερα. Σας ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ κυρία Βόρτμαν Κόλ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και την κυρία Γιαλέσεντερ για την ε, συνεργασία για να καταλήξει σε ένα καλό αποτέλεσμα αυτή η έκθεση είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε τι γίνεται και με τις θαλάσσιες μεταφορές και τους εκεί επιβάτες. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στα βασικά σημεία γιατί υπάρχουν εδώ πέρα 53 τροπολογίες που δεν νομίζω ότι θα πρέπει να σας προβληματίσουν αλλά το πρόβλημα είναι βεβαίως το πεδίο εφαρμογής και πώς θα εφαρμοστεί Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε και ο κ. Γκρός εδώ πέρα. Μιλάμε για τα δικαιώματα των επιβατών, αλλά πρέπει να είμαστε και λογικοί, να έχουμε πράγματα τα οποία θα είναι εφαρμόσιμα για τις πολλές μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εδώ πέρα. Εδώ πέρα συχνά μιλάμε για επιχειρηματίες που κυβερνούν μόνοι τους το πλοίο και δεν έχουν καν γραφείο δεν μπορούν να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις ούτε έχουν χρόνο για οτιδήποτε άλλο γιατί κυβερνούν όπως σας είπα το πλοίο τους και εδώ πέρα αυτό θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας Λέτε πως θέλουμε να δώσουμε στην εσωτερική πλοία ιδιαίτερη θέση, να είμαστε πιο ευέλικτοι και να δούμε εκεί το όριο των 36 επιβατών. Νομίζω ότι το έχουμε, έχουμε τονίσει πάρα πολύ τους 12 επιβάτες ως ε, όριο και δεν νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο ε, για τις ε, επιχειρήσεις αυτές και με 36 επιβάτες είναι σε μικρά πλοία ή σε ιστορικά πλοία τα οποία δεν είναι σε θέση να υποστούν ανακατασκευή ή τόσο μεγάλες επενδύσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως δεν θα τα βγάλουν πέρα οι επιχειρηματίες. Μην σας δώσω εδώ πέρα την εντύπωση πως δεν με ενδιαφέρουν τα δικαιώματα των επιβατών. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμένα. και πρέπει πράγματι να μπουν στην ομοθεσία, αλλά να είμαστε λίγο λογικοί. Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα από συγκεκριμένα άρθρα, να δείτε τι προτάσεις έχω κάνει. Εντάξει, μπορούμε να παραμείνουμε. Π.χ. στο σημείο 8,2 που μιλάμε για εναλλακτικέ μεταφορές, 8,5, άρθρο 15, 25 και 30. 5. Προσπαθούμε δηλαδή εδώ πέρα να δώσουμε μια σαφήνεια στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Νομίζω πως εδώ πέρα με τους 36 watts θα έρθουμε θα είναι σαφή τα πράγματα το τι μπορεί να περιμένει ο επιβάτης αν θα κατευθύνεται σε μεγάλο ε, ή μικρότερο πλοίο. Θέλουμε νομίζω να διατηρήσουμε ένα διπλό σύστημα με το κομμάτι αυτό και των 12 και μια πρόβλεψη για τα ιστορικά πλοία και τις ε, εξαιρέσεις και την ευελιξία που υπάρχει εκεί πέρα. Κατά την άποψή μου λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο, να είμαστε κάπως πιο ευέλικτοι και υπάρχει νομίζω αρκετά μεγάλη πλειοψηφία στο Συμβούλιο που το επιθυμεί αυτό. Και αυτά δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο. Συμφωνούμε εξ ονόματος ομάδας μου. Ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάου. Eh, ah. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Επιτροπής και φυσικά πρώτα απ' όλα την κυρία Γιάλα για τις τεράστιες προσπάθειες που κάνει για να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση. Δεν πρόκειται να επιμείνω διεξοδικά στα διάφορα σημεία και στις διαφωνίες μας. Τα ανέφερε η συγγήτρια. Συνεχίζονται άλλωστε οι συνομιλίες με το Συμβούλιο. Θα ήθελα να σας πω ότι ούτε για το πεδίο εφαρμογή έχουμε ακόμη συμφωνία. Εμείς προτιμούμε την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκείνη τη θέση. Ούτε συμφωνούμε με την προσωρινή εξαίρεση δύο ετών για πλοία άνω των 300 μέτρων, γιατί δημιουργεί μια βεβαιότητα και ανασφάλεια αυτό το μέτρο. Συμφωνία δεν υπάρχει ούτε και για τις αποζημιώσεις, παρόλο που υπήρξε κάποια σύγκληση. Δεν συμφωνούμε με το ανώτατο όριο του Συμβουλίου. Και παρόλο που συνεχίζουν τι διαπραγματεύσει ούτε με τη θέση σε εφαρμογή του κανονισμού αυτού συμφωνούμε. Την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ δηλαδή. Φυσικά θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες εγγύσει στους χρήστε, στους επιβάτες. Και καλό θα ήταν η απάντηση στα παράπονα να γίνεται το συντομότερο δυνατό σε μια συγκεκριμένη προθεσμία. Άσχετα από το αν γίνεται δεκτή η αιτία ή όχι. Δεν είμαστε υπέρ της, ε, του τεκμηρίου που δίνει αυτή η διοικητική σιωπή. Συμφωνούμε με την επέκταση των προδιαγραφών ποιότητα και κάτω από τις 100.000 μετακινήσεις επιβατών. Υπάρχουν πολλά θέματα λοιπόν που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασία και συζήτηση, αλλά σε ένα θέμα που διαφορούμε κάθετα με το Συμβούλιο είναι η πιθανότητα άρνησης ε, επιβίβασης σε ανθρώπους με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα όταν δικαιολογείται κάτι τέτοιο για λόγους ασφάλειας ή υγείας. Αυτό το σημείο για μας θα είναι νευραλγικό. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η ασφάλεια να είναι λόγος για άρνηση επιβίβασης ε, ή υγεία. Μάλιστα για ένα όριστο κριτήριο γιατί δεν προσδιορίζεται ποιος έχει δυνατότητα να πετήσει ή να εγκρίνει κάτι τέτοιο. Συμφωνούμε ριζικά ε, διαφωνούμε ριζικά με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό και είναι θέμα κλειδί για την ομάδα μα. Θέλουμε να προστατεύσουμε του επιβάτε και τα δικαιώματά του, αλλά να προστατεύσουμε και αυτού που έχουν αναπηρίε ή περιορισμένη κινητικότητα. Μάλιστα, μην ξεχνάτε ότι όλοι μα είμαστε ε, δυνάμοι άνθρωποι με αναπηρίε ή με περιορισμένη κινητικότητα και όλοι εδώ οι παρόντε, α μην το ξεχνάμε λοιπόν. Η ομάδα μας, οι φιλελεύθεροι, θα υποβάλουμε και άλλες τροπολογίες γιατί είμαστε διαθέσιμοι να καταλήξουμε στη συμφωνία και πιστεύουμε ότι μπορούμε και να το κάνουμε. Κυρία Λίχτεμπεργκερ. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι την ίδια συζήτηση έχουμε εδώ πέρα που είχαμε και με τα λεωφορεία. Δηλαδή δίνουμε δικαιώματα στους ανθρώπους με κινητικότητα όταν είναι εύκολα, όταν είναι πιο δύσκολα καλύτερα λέμε όχι. Οπότε κάποια από τα επιχειρήματα τα οποία ακούστηκαν δεν ξέρω μου ακούγονται λίγο περίεργα. Να αναφερθώ λοιπόν σε αυτά. Πρώτα απ' όλα το θέμα του μεγέθους 12 ή 36 άτομα. Πρέπει να αποφύγουμε να κατέβουμε νομίζω κάτω από αυτό το όριο για να βελτιωθεί η κατάσταση. Δεύτερον, τα ιστορικά πλοία. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει μετασκευή. Αλλά φοβάμαι ότι μετά οτιδήποτε είναι παλαιότερο από 10 χρόνια θα γίνει αυτομάτως ιστορικό και θα έχουν όλη εξαίρεση και δικαιολογία. Ε, ε, δεν είναι θέμα μόνο μετασκευής, που δεν είναι και τόσο τραγική. Δεν μιλάμε εδώ πέρα μόνο για όσους ε, έχουν ένα πυρικό καροτσάκι, έχουν ανθρώπους που δεν βλέπουν καλά, δεν ακούνε καλά. Δηλαδή τα πολλά, δεν χρειάζονται, τα πολλά πράγματα δεν χρειάζονται και μεγάλες μετασκευές, χρειάζονται μόνο τη θέληση να κάνουμε κάτι ε, για αυτούς τους ανθρώπους. Και κάτι άλλο το οποίο μου φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, το έχω συζητήσει με την κυρία Γιαλασέντερ τα λιμάνια. Δηλαδή, αν δεν τα καταφέρουμε και στα λιμάνια να υπάρχει προσβασιμότητα, ε, δεν μπορούμε να αναμένουμε άτομα με κινητικές δυσκολίες ή με καροτσάκια ε, πώς θα, θα και θα βρεθούν στο πλοίο. Από το αυτοκίνητο ως διαμαγείας πρέπει και το λιμάνι να δίνει την δυνατότητα να έχει δηλαδή αυτές τις ανάλογες υπηρεσίε όπως υπάρχουν στα αεροδρόμια. Βεβαίω, εντάξει, μπορούμε να πούμε 100 φορές ε, ναι, εντάξει, μικρή επιχείρηση κινδυνεύει. Γιατί δεν υπάρχουν στηρίξεις, ε, επιδοτήσεις για την εφαρμογή αυτών των πραγμάτων μια οικονομική βοήθεια από πλευράς των κρατών. Επενδύουν πάρα πολλά στις υποδομές. Με κάποιες μετασκευές. Ε, και με αυτές θα απασχοληθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό δημιουργεί θέσεις εργασίας και αυτό προωθεί την οικονομία. Απλά πρέπει να το αντιληφθούμε ως τέτοιο. Αυτό είναι όλο. Εγώ είμαι βαθύτατα πεπισμένη πως ε, μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα ένα πολύ σημαντικό βήμα. Τέλος, για την ανεξάρτητη υπηρεσία. Έγινε αποδεκτή, χαίρομαι, γιατί αν δεν έχουμε μια ανεξάρτητη υπηρεσία στην οποία μπορεί να στραφεί κανείς όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά του, τότε θα σταματήσει όλη η υπόθεση πριν καν ξεκινήσει. Ελπίζω λοιπόν και εδώ πέρα να έχουμε σύντομες μεταβατικές προθεσμίες. Ελπίζω εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Ένωση να μπορέσουμε να πούμε πως ναι η σύμβαση για τα δικαιώματα των αναπήρων είναι κάτι που παίρνουμε σοβαρά και θέλουμε να τους κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη. Απευθύνω έκκληση λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, μην χάσουμε αυτόν τον στόχο. Ξέρετε πως και εγώ είμαι υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά δεν μπορεί να είναι μονίμως η δικαιολογία μας για α, όταν θέλουμε να λάβουμε κάποια μέτρα για την κινητικότητα. Ας μην το κάνουμε αυτό. Ούτε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή ούτε αυτές ε, βοηθάμε έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σχετικά σύντομη γιατί ήδη ακούστηκαν αρκετά πράγματα. Να υπενθυμίσω δύο πραγματάκια που αναφέρθηκαν ήδη. Πρώτα απ' όλα η υγειονομική λόγη για την πρόσβαση, κύριε Βιβάρου το είπε ήδη για την Άλντε πως δεν είναι αποδεκτό αυτό. Πρέπει να εξηγήσουμε τι εννοούμε εδώ πέρα, γιατί οι λόγοι υγείας μόνο δεν, δεν νομίζω να μπορεί να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο. Δεύτερον, να λάβουμε υπόψη πράγματι το εάν ε, γίνεται κάτι τέτοιο στην πράξη. Σύντομα τώρα, για τα ιστορικά ε, πλοία. Εγώ έχω πάει και σε ιστορικό ιστιοφόρο. Μπορούν να ανέβουν πάνω άνθρωποι με ε, καροτσάκι. Απλά δεν μπορούν να κατέβουν κάτω από το κατάστρωμα. Αυτό είναι δύσκολο. Επίση, δεν είναι έτσι τόσο απλό να έγιναν αυτέ οι μετασκευέ με όλη την καλή θέληση που μπορεί να έχει κανείς. Να δούμε δηλαδή το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται. Και τέλο μετά να δούμε πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι να κατέβουν κάτω στα, από το κατάστρωμα στα υπόλοιπα καταστρώματα. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ. Κυρία Γέγκερ από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν θα ήθελε να συγχαρεί την κυρία Γιάλα Σέντερ, την εισηγήτρια, και τους κοιόδες εισηγητές για τη σκληρή δουλειά που κατέβαλαν για αυτό το φάκελο. Με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι όλοι προσπαθούν να επιτευχθεί συμφωνία, ε, που, κάτι που είναι πολύ θετικό και για τους επιβάτες αλλά και για τη βιομηχανία. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής για την υγεία, για τις αποζημιώσεις, ε, επιπρόσθετη αποζημίωση σε σχέση με την τιμή του εισιτηρίου, αλλά πιστεύουμε ότι τελικά θα βρεθεί συμφωνία. Για το πεδίο εφαρμογή, θα ήθελα να τονίσω ότι συμφωνούμε με κάποιους ε, τους ε, ομιλητές ότι πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα κριτήρια και το διπλό κατόφλι θα δημιουργήσει σύγχυση στους επιβάτες. Απ' την άλλη όμως πιστεύουμε ότι μπορεί να βρεθεί συμβιβασμός μεταξύ του 36 και του 12 της αρχικής πρότασης της Κομισιόν. Και πιστεύουμε ότι κάποια σκάφη ήδη αποκλείονται. Ε, μην ξεχνάτε ότι ο ορισμός αφορά ε, πλοία μέχρι 500 μέτρα ή μέχρι 3, μέτρα, 3 ε, άτομα πλήρωμα. Ο συμβασμός είναι κάπου εκεί, κάπου στο μεταξύ. Οι επιβάτες της θαλάσσιας μεταφορές έχουν ε, περιμένουν εδώ και χρόνια για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε περαιτέρω. Η Κομισιόν θέλει να διευκολύνει την επίτευξη συμβιβασμού που θα επιτρέπει μια συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση για το καλό των επιβατών των θαλασσιών μεταφορών. Η κυρία Γιαλασέντε. Eh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους. Και το παιδί εφαρμογή, όπως είπε η κυρία Γέγκερ και άλλοι συνάδελφοι, θα το διαπραγματευτούμε και πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη σύγκληση απόψε με το Συμβούλιο. Άλλωστε το δέχεται αυτό και ο κλάδος. Για το θέμα των αποζημιώσεων υπάρχει θέμα περιθωρίου και το θέμα της υγείας είναι ακόμη πιο περίπλοκο. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή σε ένα τόσο περίπλοκο κλάδο όπως είναι οι ναυτιλιακές μεταφορές για να ξεκινήσουμε μια τέτοια συζήτηση. Αναγνωρίζω τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλει η Ισπανική Προεδρία για την ε, προσέγγιση του Συμβουλίου στη θέση του Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι αυτά τα τρία σημεία είναι τα πλέον επίμαχα και τα πιο περίπλοκα, αλλά ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Τουλάχιστον θα τα αφήσουμε εκρεμή εν αναμονή μια συμπερίληψή του στο μέλλον. Για τα υπόλοιπα σημεία ήδη υπήρξε σημαντική σύγκληση και η εκπεφρασμένη βούληση να καταλήξουμε σε συμφωνία από την πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βοήθειά της. Ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 6η Μαΐου και όπως και για το προηγούμενο θέμα 1η Ιουνίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και θα ψηφίσει η Ολομέλεια τον Ιούλιο. Ε, έχουμε την 6η Μαΐου την καταληκτική ημερομηνία για τις οπολογίες αυτής της έκθεσης και για την έκθεση του κ. Καντσάν ε, την 7η Μαΐου. Πάμε τώρα ε, στην επόμενη έκθεση του κ. Μαρινέσκου, Ευρωπαϊκό Συνδρομικό Δίκτυο. Κύριε Μαρινέσκου. Αγαπητοί συνάδελφοι, από τελευταία φορά που συζητήσαμε αυτό τον κανονισμό, Είχα συναντήσεις με τους κοιόδης εισηγητές. Θέλω να τους ευχαριστήσω πραγματικά για τη συνεργασία και για τη διαθεσιμότητά τους. Επίσης είχαμε και μια συνάντηση τριμερούς διαλόγου με το Συμβούλιο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι λοιπόν. Μια σειρά προφορικών τροπολογιών στη θέση που έχω ήδη υποβάλει. Θα, προσπαθώ, θα προσπαθήσω να τις παρουσιάσω αυτές τις προφορικές τροπολογίες και να σας πω τι συζήτησα με το Συμβούλιο και τους κοιόδη συζητητές και πού επιτύχαμε συμφωνία. Συζητήσαμε επίσης ξανά μετά από κάποιες προτάσεις που έκανα για συμβαστικές τροπολογίες ε, συζητήσαμε με τους κοιόδης συζητητές και συμφωνήσαμε. Θα, ε, ε, θα, ξέρετε, θα ότι υπήρχαν 80 τροπολογίες. Κατάφερα μέχρι στιγμής να τις συμπεριλάβω όλες στους συμβιβασμούς ή σε άλλου τύπου τροπολογίες. Προκειμένου να συμφωνήσουν τελικά έτσι οι πολιτικές ομάδες. Να αναφέρω και κάτι άλλο δύο σημαντικά πράγματα κατά την άποψή μου. Καταρχάς, δέχτηκα την θέση του Συμβουλίου, ε, τη συμπερίληψη δηλαδή ενός και την έγκριση διαφόρων διαδρόμων μέσω αυτού του κανονισμού. Έχουμε ένα αρχικό ανταγωνιστικό δίκτυο τέτοιων μεταφορών εμπορευμάτων και προσθέτουμε τώρα και αυτούς τους ε, διαδρόμους. Θα πρέπει να συζητήσουμε βέβαια από ποιες πόλεις ε, περνάνε αυτοί οι διάδρομοι, αλλά ελπίζω να το συμφωνήσουμε τελικά αυτό το θέμα για τους διαδρόμους. Δεύτερον, ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκε είναι το one-stop shop, το λεγόμενο. Νομίζω ότι συμφώνησαν από αυτού τώρα οι πολιτικές ομάδες και το Συμβούλιο. Γι' αυτό το πολύ σημαντικό θέμα είναι πολύ σημαντικό οι χρήστες των εμπορευματικών διαδρόμων να απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε ένα μόνο συγκεκριμένο σημείο και να λαμβάνουν μία έγκριση για τη διαδρομή. Για τις διαπραγματεύσεις ε, με το Συμβούλιο υπάρχει ένα θέμα που είναι ακόμα επίμαχο. Οι εγκεκριμένοι ετούντες Ίσως εδώ έχουμε πρόβλημα με το Συμβούλιο. Μα ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ αυτό το θέμα, όπως θα δείτε και από τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Θέλουμε ανοιχτή αγορά και θέλουμε να παραμείνει αυτή η ανοιχτή αγορά στην Ευρώπη. Αλλά το Συμβούλιο δεν έχει συμφωνήσει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα πρέπει να δούμε εάν τελικά θα συμφωνήσουμε το Συμβούλιο για αυτό το σημείο ή όχι. Περιμένω τις απόψεις σας σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που έχω υποβάλει και την πρόταση με τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Μετά από τις σημερινές συζητήσεις με τους ε, σκιώδεις εισηγητές, θα κάνω κάποιες αλλαγές στον κατάλογο των ψηφοφοριών εν ευθέτω χρόνο και θα σας τον υποβάλω για να τον εξετάσετε, ούτως ώστε να είστε έτοιμοι για την αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Θα ακούσουμε τους σκιώδεις εισηγητές και πρώτα απ' όλα τον κύριο Λιμπεράτσκι από τους ε, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτά που μας είπε ο εισηγητής μας ο κύριος Μαρινέσκου. Βέβαια, οι τροπολογίες και οι δικές του, αλλά και των άλλων βουλευτών, τις αναλύσαμε. Όπου υπήρξε συμφωνία, το διαπιστώσαμε όπου υπήρξε διαφωνία, επίσης το αναγνωρίσαμε, γι' αυτό και θα υποβληθούν κάποιες συμβεβαστικές τροπολογίες, είτε προφορικές είτε γραπτές, για τη σύγκληση των απόψεων. Θα ήθελα πάντως να επισημάνω ότι στη δική μου ε, πολιτική ομάδα ξεκινήσαμε με την προϋπόθεση ότι όλοι συμφωνούμε με την ιδέα μια, ενός ανοιχτού ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Βέβαια, στις διάφορες φάσεις της συζήτησης σκεφτήκαμε πως θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιό της και να μας υποβάλει ένα νέο. Παρ' όλα αυτά τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε σημαντική πρόοδο σε μεγάλο βαθμό χάρη και στην ιόβη υπομονή του κυρίου Μαρινέσκου γιατί άκουγε υπομονετικά και στοικά τις ε, θέσεις του Συμβουλίου και τις ε, των διαδοχικών προεδριών. Και δικαιώθηκε και ο πρόεδρος μας, ο Μπράιν Σίμψον, που είπε ότι οι σιδηροδρομικοί πάντοτε θα βρίσκουν λόγους για να αντισταθούν σε κάτι που θα μας πλησιάσει σε μια ε, εύρυθμη, αποτελεσματική και δίκαιη σιδηροδρομική αγορά. Τώρα βέβαια δεν έχουμε 180 λόγους των σιδηροδρομικών, αλλά 127. Αλλά είναι εύκολο να βρεθούν φράγμοι και περιορισμοί. Το πιο σημαντικό πάντως είναι ο ορισμός του διαδρόμου μεταφοράς. Τελικά είδαμε ότι των δημιουργίων πνευματικών διαδρόμων είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε αυτό το θέμα, αλλά και το θέμα της σύνδεσης. Όχι μόνο τη δημιουργία εμπορευματικών διαδρόμων, αλλά και το θέμα της σύνδεσης βορανότου, για παράδειγμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μετά από εκτενείς συζητήσεις και εξετάσεις, καταλήξαμε στην πρόταση του One Stop Shop. Και νομίζω ότι εκεί έχουμε συμβαστική λύση και μπορούμε να έχουμε γιατί για κάθε τέτοιο διάδρομο τέτοιο one-stop shop. Βέβαια εδώ υπάρχει πρόβλημα με, την, με τους διαχειριστές των δίκτυων της υποδομής και τους εταίρους μας. Τους διαχειριστές δηλαδή των δικτύων. Πάντως υπάρχει και το θέμα της επίλυσης των διαφορών και για το One Stop Shop αλλά και για το ποιες χώρες ενδιαφέρονται και θα συνδεθούν με αυτές τους εμπορευματικούς διαδρόμους. Και φαίνεται ότι με εξαίρεση τη Μάλτα και την Κύπρο ε, δεν ε, αφήσαμε κανένα, καμία χώρα απ' έξω σε ό,τι αφορά το χάραξη αυτό το, αυτούς ε, τους εμπορευματικούς διαδρόμους. Μέχρι και τη Σλοβενία τελικά την συμπεριλάβαμε. Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις που τις συμμεριζόμαστε και εμείς. Για παράδειγμα, ο αρχικός ενθουσιασμός έχει μετριαστεί κάπως ό,τι αφορά τη δημιουργία τέτοιων εμπορευματικών διαδρόμων. Και Μερικοί δεν θέλησαν να συμπεριληφθούν σε αυτούς τους διαδρόμους, γιατί σκέφτηκα τις ευθύνε που θα συνδεθούν με τέτοια συμμετοχή σε σιδηροδρομικούς διαδρόμους. Επίσης και οι προθεσμίε που προτείνονται, δηλαδή τα δύο χρόνια, έξι μήνες για την υποβολή καταλόγων συνδέσεων, η προσφορά, η ικανότητα των μεταφορέων για τη δυνατότητα χορηγήση ε, σλότ χρονοδιαδρόμων για τις εμπορευματικέ μεταφορές. Αυτά τα σημεία είναι αρκετά επίμαχα, αλλά μετά από συζήτηση βρέθηκε κάποια συμφωνία και η δική μου πολιτική ομάδα είναι αρκετά ικανοποιημένη. Γιατί από την αρχική άρνηση της πρώτης ανάγνωσης κάναμε ένα κύκλο σχεδόν και δεχτήκαμε τελικά την κοινή θέση και υπήρξε σημαντική διαφορά. Έχουμε συντάξει ένα κατάλογο ψηφοφορίας που είναι συνενετικός. Έχουμε και κατάλογο ψηφοφορίας στον οποίο θα συγκεντρώσουμε σημαντική πλειοψηφία πιστεύω και θα ήθελα να αποτανθώ στους συναδέλφους και τις συναδέλφιες και να πω ότι σε πολλές περιπτώσεις θα χρειαστεί να μετριάσουμε τις φιλοδοξίες μας και να παραιτηθούμε από αυτές. και ίσω χρειαστεί να αποσύρουμε και ορισμένε τροπολογίε Και εγώ από έσυρα κάποιε τροπολογίε το ίδιο και ο κύριο Μαρινέσκου. Μην θεωρείτε λοιπόν ο ΣΥΤΑ να δεν γίνει δεκτή κάποια, κάποια τροπολογία σας, γιατί η επιτυχία θα κριθεί από το αν θα εγκρίνουμε το συνολικό σχέδιο και θα βοηθήσουμε τους σιδηροδρομικούς ε, να προσαρμοστούν σε αυτή την κατάσταση της ε, κρίσης και να σηκώσουν το κεφάλι και να ακολουθήσουν και αυτό το δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπιλμπά από τους Φιλελεύθερους. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μαρινέσκου γιατί σας διαβεβαιώ ότι καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και μαζί του υποφέρουν και οι βοηθοί και η γραμματεία πολύ περισσότερο από μας. Το πρωί μάλιστα είχαμε μια τελευταία συνεδρίαση, υπεβάλαμε όλες τις τροπολογίες μας και οι φιλελεύθεροι κατέθεσαν πολλές τροπολογίες που δεν είχαν αρχικά γίνει δεκτές στις προηγούμενες ε, διαπραγματεύσεις. Εμείς σταχθήκαμε υπέρ της ε, πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της θέσης της πρώτης ανάγνωσης και αυτήν ε, προασπίσαμε και σε όλες τις συζητήσεις παρόλα αυτά συμμετείχαμε με διαλλακτικό πνεύμα, με στόχο την διαμόρφωση ενός οριστικού σχεδίου που θα έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Και προσπαθήσαμε να υπερασπίσουμε υπό αυτό το πρίσμα της τροπολογίας μας, υπό το ευρωπαϊκό δηλαδή πρίσμα. Πολλές δυσκολίες αντιμετώπισε αυτό το σχέδιο και ο αρχικός ορισμός του, του Συμβουλίου μεταξύ του πρώτου παραρτήματος όπου θα περιλαμβάνονταν τα τα... οι προϋποθέσεις για τους νέους ε, διαδρόμους τελικά καταφέραμε το παράρτημα 2 να συμπεριληφθεί στο διατακτικό του κανονισμού και εκεί συγκεντρώσαμε ευρεία συμφωνία. Το παράρτημα 1 αναφέρει τους διάφορους διαδρόμους Και μάλιστα πολλές φορές ρωτήσαμε το Συμβούλιο. Γιατί έγινε η πρόταση για του συγκεκριμένου διαδρόμου και όχι για άλλου, για παράδειγμα. Δυστυχώ δεν έλαβα ικανοποιητική απάντηση από το Συμβούλιο. Η μόνη απάντηση που έλαβα ότι αυτή είναι η απόφαση των α, χωρών. Ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα αλλάξει αυτή η συμφωνία και γι' αυτό η τροπολογία μας ως προς το παράρτημα 1 θα καταψηφιστεί για να είμαστε συνεπείς με την αρχική μας θέση, αλλά θα υποστηρίξουμε τις υπόλοιπες τροπολογίες που αφορούν τους διαδρόμους. Επαναλαμβάνω, εμείς μένουμε πιστοί στη θέση του Συμβουλίου της πρώτης ανάγνωσης. Σήμερα το πρωί παρόλα αυτά κάναμε πολλές, ε, πολλούς συμβιβασμούς. Αυτό που μας ανησυχεί πάρα πολύ είναι το θέμα του One Stop, της ενιαίας θηρίδας. Υπάρχουν εκεί τρεις διαφορετικές θέσεις. Η τρίτη ανέκυψε από την σημερινή συζήτηση η μία πρόταση μιλάει για one-stop, μια νέα θηρίδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλους τους διαδρόμους. Φαίνεται ότι αυτή μάλλον δεν θα ευοδοθεί, δεν θα τελεσφορήσει. Η δεύτερη πρόταση είναι ενιαία θηρίδα εθνική, για κάθε χώρα δηλαδή. Και μάλιστα σήμερα από τη συζήτηση προέκυψε και το πρότεινα και εγώ στην ε, κοινοβουλευτική ομάδα, είναι να υποβάλουμε μια τρίτη εναλλακτική λύση που να μην είναι προσωπική πρόταση καθενός, αλλά θα μπορούσε να είναι κοινή λύση, δηλαδή μια ενιαία θηρίδα για κάθε διάδρομο. Ούτε για κάθε χώρα, ούτε για ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι θα έχουμε και μια ευρωπαϊκή διάσταση σε αυτό το σχέδιο. Θα μπορέσουν και τα κράτη-μέλη να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να λειτουργήσουν αυτοί οι διάδρομοι μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της ανέβρεσης κοινών λύσεων με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και πιστεύω ότι αυτή η λύση θα μας βοηθήσει να φτάσουμε και σε συμφωνία για το σχέδιο αυτό. Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό των επενδύσεων, παρά την αρχική διστακτικότητα του Συμβουλίου να καλύψει και το θέμα αυτό, τελικά συμπεριλήφθηκε κάποιο σημείο και μας ικανοποιεί η μνή αυτή του προγραμματισμού των επενδύσεων κατά την εκτέλεση των σχεδίων. Γενικώ πάντως και μετά από την εξέταση και αυτών των πιο επιμαχών σημείων ευελπιστώ ότι αύριο στην ψηφοφορία θα καταλήξουμε στη συμφωνία και θα καταλήξουμε σε ένα σχέδιο που θα μοιάζει περισσότερο με την, θέση, την κοινή θέση του, Συμβουλίου στην πρώτη, του Κοινοβουλίου συγγνώμη, στην πρώτη ανάγνωση. Ο κύριος Κράμερ για τους πράσινους. Ναι. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον συγητή και τη γραμματεία που μας στήριξε και τους κοιόδης συγητές. Δύο ουσιαστικά θέματα ήταν για μας αποφασιστικά για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν να υπάρξει ένα δίκτυο μεταφοράς εμπορευμάτων κατά προτεραιότητα στην Ευρώπη χωρίς να μας απασχολούν ε, οι ζημίες Κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι από την Γερμανία και εκεί πέρα σε όλους ε, τους ε, σύρμους ε, είναι μικτές οι μεταφορές. Υπάρχει ένα πολύ καλό δίκτυο βέβαιος ΤΖΒ, αλλά τα υπόλοιπα τρένα είναι όλα μεικτά, οπότε θέλουμε να υπάρχει μια γενική μια γενική φύλαξη αν θέλετε, μια κράτηση των ε, διαδρομών αυτών ε, για να μπορούν να περνάνε αυτά τα εμπορευματικά τρένα και να μην ε, Να μην σημαίνει αυτό βεβαίω πώ θα καταργηθούν τα μικρά περιφερειακά τρένα, γιατί δεν μπορούμε εμεί να πούμε Α, τώρα έχουμε ένα ωραιότατο δίκτυο μεταφορά εμπορευμάτων, οπότε θα πρέπει να καθυστερήσει το τρένο σα εδώ πέρα τη τοπική συγκοινωνία. Αλλά να υπενθυμίσω κάποια πράγματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για εμά. Μιλάμε για τι πράξει αυτέ κατεξοδότηση που εμφανίζονται τώρα. Είναι σαφέ εδώ πέρα πώ θα συμμετάσχει το Κοινοβούλιο. Πως η Κομισιόν δεν έχει το δικαίωμα να κάνει μόνη τη αλλαγές, αλλά δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε μόνο, χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη μας εάν είναι να αλλάξει κάτι. Και πράγματι έτσι πρέπει να γίνει. Δεύτερον, τι θα κάνουμε με αυτό το One Stop Shop και τα διάφορα διαφορούς φορείς εκεί πέρα, όταν αυτά τα δύο διαφορούν μεταξύ τους για την διαχείριση των υποδομών. Είναι σαφές πως η απελευθέρωση αυτών των δικτύων θα πρέπει να είναι ε, και η διαχείριση βεβαίως στο εθνικό δίκτυο. Δεν μπορεί να πει δηλαδή η υπερεθνική αρχή ότι αυτό δίκτυο τώρα το διαχειριζόμαστε εμείς και θα κάνετε εσείς με τις δικές συγκοινωνίες αδιαφορούμε. Δεν γίνεται αλλά εάν ε, ανοίγει το δίκτυο από τους ε, διαχειριστές ε, αυτούς των υποδομών, τότε να πούμε ναι εντάξει έτσι θα γίνει η κυκλοφορία γιατί αυτή είναι η ανάγκη. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως πριμοδοτούμε. δηλαδή επίσης Όταν λένε πως το δίκτυο εκείνες ώρες είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτό. Δεν μπορούμε μετά να το πάρουν πίσω ε, όταν βλέπουν ότι έχει ανταγωνιστής, γιατί κάποιοι μπλοκάρουν ε, ε, και εθνικές επιχειρήσεις σιδηροδρόμου μπλοκάρουν 20-30 δρομολόγια μόνο και μόνο για να μην πάει κάποιος ανταγωνιστής και τα χρησιμοποιήσει. Εμείς θέλουμε όμως περισσότερη κυκλοφορία σιδηροδρομικές γραμμές και όχι μόνο ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα γιατί έτσι που θα καταλήξει η κίνηση θα πάει στους δρόμους. Αλλά εάν στο διάδρομο βλέπουμε πως εκεί και εκεί υπάρχει η ελεύθερη γραμμή έτσι πρέπει να γίνεται. Τώρα για το One Stop Shop. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλά πράγματα. Τι ήταν η δική μας ιδέα πως πρέπει να υπάρχει μία αρχή έτσι ώστε όταν μία επιχείρηση ζητάει ένα κομμάτι της γραμμής να είναι ανοιχτό να μην χρειάζεται να κάνει τέσσερις αιτήσει σε τέσσερις διαφορετικούς διαχειριστές των υποδομών να υπάρχει μία απόφαση να απευθύνεται σε έναν και να τελειώνει εκεί πέρα. Αλλά βεβαίω υπάρχει ένα ανοιχτό ε, ερώτημα. Το Συμβούλιο Μιλάει σαν να υπάρχουν δύο αρχές, μία δηλαδή για να συγκεντρώνει και να εξετάζει τις αιτήσει και άλλη μία είναι υπεύθυνη για τις μεσομακροπρόθεσμες ε, επενδύσεις. Το να τις χωρίσουμε αυτές ε, σημαίνει μόνο μία διπλή συζήτηση. Εάν υπάρχει κάπου μεγάλη σύντηση και δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί 5-6 χιλιόμετρα δεν υπάρχει μια διπλή ή τριπλή γραμμή, εάν τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά, τότε να ληφθεί και η απόφαση ναι να το κάνουμε το επόμενο χρόνο. Βεβαίω εντάξει χρειάζονται περισσότερη μηχανική, αλλά ίσω να, να γίνεται. Να μπει μια δεύτερη γραμμή όπω π.χ. στο, στο λιμάνι του, του Ροστόκ που χρειάστηκαν 60 χρόνια και Μπολόνια Βερόνα επίσης ε, σχεδόν κράτησε 100 χρόνια αλλά ελπίζω να αλλάξει κάτι. Οπότε να φύγουν από τη μέση αυτές οι προτεραιότητες και οι κρατήσεις των γραμμών. Βρήκαμε νομίζω συμβαστικές ε, λύσεις, οπότε θέλω να ευχαριστήσω εδώ πέρα όλες, ε, όλους τους συναδέλφους. Βλέπω και το σφυράκι του Προέδρου, οπότε τελειώνω. Thank you for the Κύριος Έπι, από τους ε, συντηρητικούς. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Και εγώ υποστηρίζω σε γενικές γραμμές την έκθεση και τους συμβιβασμούς που έχει προτείνει ο εισηγητής. Συμφωνώ κυρίως με την αρχή των διαδρόμων. Το μόνο ερώτημα είναι το αν θα λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία. Πρέπει να το διαρωτηθούμε αυτό ως Ευρωπαίοι. Θα δημιουργήσουμε ένα κοινό φορέα και αυτή την ενιαία θηρίδα, η οποία, διαρωτώ θα λειτουργήσει. Δεν θα ήταν καλύτερο να κρατήσουμε το σύστημα των εθνικών φορέων υποδομών για ένα χρονικό διάστημα. Ε, απλώς να διασυνδέονται καλύτερα και να έχουμε ένα ρυθμιστικό σύστημα που ε, εξετάζει τις προθεσμίες, τη διαφάνεια κτλ. Γιατί αν αυτό το σύστημα της ενίας τρίδας δεν λειτουργήσει, δεν θα έχουμε τίποτα. Θα περιμένουμε μονίμως ε, τους χρονοδιαδρόμους και θα έχουμε μονίμως καθυστερήσεις. Υπάρχουν μεγάλες χώρες και πολύ πυκνές χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία. Ε, δεν μπορεί μια τέτοια θερίδα πάντα να αποφασίζει αν θα περάσει το, το τρένο ξέρω από την τάδε πόλη, τη δίνα πόλη. Χρειάζεται συνεργασία. Συμβιβαστικά λοιπόν θα έλεγα καλύτερα να διασυνδεθούν καλύτερα για κάνα δύο χρόνια τα συστήματα που υπάρχουν ήδη και μετά να κάνουμε μια αξιολόγηση για το αν μπορούμε να έχουμε αυτή την ενιαία θηρίδα. Να έχουμε δηλαδή μια πιο α, βαθμιαία προσέγγιση. Ε, θα θυμάστε τι κάναμε με το ταχυδρομικό τομέα. Ε, όταν ξεκινήσαμε πριν 10 χρόνια, ας πούμε, είχαμε αντιδιαμετρικές απόψεις πρώτα, θα το θυμάστε. Αλλά τελικά βαθμιαία, ας πούμε, πλησιάσαμε ο ένας τον άλλον. Νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν και εδώ να είχαμε μια πιο βαθμία προσέγγιση παρά να επιβάλλουμε μόνο αυτή την ε, νέα θηρίδα. Γι' αυτό λοιπόν θα απέχω. Ο κύριος Ράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και να πω εξ ονόματος του ΕΛΚ πως βεβαίως εντάξει είναι σημαντικό να υπάρχει εδώ πέρα πράγματι μια ευρωπαϊκή διάσταση και όχι απλή πρόσθεση εθνικών διαστάσεων, κάτι το οποίο δεν θα είναι βεβαίως τόσο εύκολο, αλλά νομίζω πως ο εισηγητής εδώ πέρα με τους κοιόδης ε, τα κατάφερε. Και δεύτερον, πράγματι πρέπει να πάμε προς αυτή την ε, κατεύθυνση. ιδέα αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει αυτόν τον υπερεθνικό και όχι έναν επιπρόσθετο χαρακτήρα όσον αφορά δε τον προγραμματισμό. Συμφωνούμε, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μακροπρόθεσμου ε, προγραμματισμού και να αντιμετωπίσουμε βραχυπρόθεσμα ιδιαίτερε καταστάσεις όταν μιλάμε για πάρα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα προγραμματισμού και για αυτές τις περιπτώσεις πράγματι πρέπει να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτεραιότητα. Με πάση περιπτώσει, ο εισηγητής ε, και όλοι όσοι εργάστηκαν εδώ πέρα έχουν την στήριξή μας και νομίζω πως θα μπορέσουμε να πείσουμε και το Συμβούλιο και την Κομισιόν να κινηθεί εδώ πέρα μαζί μας και να συνεργαστούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Αλχαντραουή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή εντάξει, τελικά είμαστε κάπως ε, πιο μακριά από ό,τι φοβόμασταν κάποιες στιγμές, αλλά πρέπει νομίζω να θέσουμε ορισμένα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, σημαίνει πρόοδο αυτός ο κανονισμός για το πώς δηλαδή θα γίνει πιο αξιόπιστος και πιο ελκυστικός ο σιδηρόδρομος. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα, η μέθοδος εάν δηλαδή η προτινόμενη λύση είναι ρεαλιστική και απλή και ευέλικτη. Και νομίζω πως μπορούμε να απαντήσουμε μάλλον θετικά, παρά το ότι τα πράγματα δεν είναι τέλεια. Δύο στοιχεία είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα ο ορισμός του σιδηροδρομικού διαδρόμου. Πραγματι εδώ στο παράδειγμα υπάρχει ένα σχετικό κατάλογος, αλλά πρέπει να υπάρχει αρκετή ευελιξία έτσι ώστε μέσω των πράξεων κατεξιοδότηση να μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα στο μέλλον και να αναμειγνύεται και το Κοινοβούλιο δεύτερον το γνωστό One Stop Shop για να υπάρξει η δυνατότητα να δημιουργηθεί αυτή η απαραίτητη υποδομή. Τώρα το να έχουμε εθνικά one stop shop δεν νομίζω ότι ευθυγραμμίζεται με αυτό το οποίο θέμε, δηλαδή μπορεί να διαλέγει κανείς νομίζω το ανάλογο σώπανα διάδρομο είναι το καλύτερο. Τώρα το υπάρχον σύστημα συντονισμού νομίζω μπορεί να ενσωματωθεί εδώ πέρα αυτό το οποίο υπάρχει τώρα. τα πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση περιπτώσει το One Stop Shop. Επίσης πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία για να δούμε τι θα γίνει με τυχόν προβλήματα, διαφορές, ε, συγκρούσεις ας πούμε, αλλά ταυτόχρονα και τελειώνω κύριε Πρόεδρε να μην δώσουμε την εντύπωση πως ε, μόνο με αυτή την νομοθεσία ως διαμαγείας θα έχουμε καλύτερες μεταφορές. Είναι ένα μέτρο μεταξύ πολλών άλλων. και πρέπει βέβαια να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στην έκθεση του συναδέλφου Γκρός για να γίνουν πιο αποτελεσματικές συνδρομικές μεταφορές και μεταφορές εμπορευμάτων ειδικότερα αλλά είναι ένα μικρό βήμα πρόοδου αυτό εδώ πάντως ο εισηγητής έχει την πλήρη στήριξή μας Ευχαριστώ η κυρία Μάισνερ συμφωνώ πλήρως με τον συνάδελφο. Είπε πως είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την μεταφορά αγαθών, αλλά όχι οπωσδήποτε το τελευταίο και το οριστικό. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Θέλουμε να λειτουργούν αυτές οι μεταφορές όπως είναι στα χαρτιά, αλλά βεβαίω όχι στην πραγματικότητα. Θα ήθελα εγώ τώρα να αναφερθώ σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Κράμερα ανέφερε πως στη Γερμανία έχουμε το πρόβλημα πως ε, δεν μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα στα αγαθά γιατί υπάρχει και η μεταφορά των προσώπων και δεύτερον βεβαίως το One Stop Shop ε, όντως στην δική μου ομάδα συζητάμε ε, μέχρι τελευταία στιγμή ποια είναι η καλύτερη λύση η κυρία Μπιλμπάου ε, έδειξε πως υπάρχουν τρεις διαφορετικές ε, λύσεις. Η πιο ευρωπαϊκή είναι να πούμε ίσως πως να έχουμε ένα one-stop shop ανά διάδρομο και να δούμε τι θα γίνει με τις εθνικές υπηρεσίες. Και εδώ πέρα συμφωνούμε με αυτό. Νομίζω τα εθνικά one-stop shop ε, δεν συντονίζονται ακόμα αρκετά καλά μεταξύ τους, αλλά δεν ξέρω εάν θα μπορούσαμε να τους υποχρεώσουμε να συντονιστούν καλύτερα, αν είναι καλύτερο αυτό, από το να κάνουμε άλλο ένα σύστημα, που σημαίνει διπλό σύστημα. Γιατί υποτίθεται ότι η Ευρώπη είναι υπέρ της απλοποίησης και όχι να γίνονται τα πράγματα πιο πολύπλοκα για να λειτουργεί έτσι το σύστημα άψογα. Οπότε συμφωνώ με όσους λένε πως θέμε ένα one-stop shop αναδιάδρομο, αλλά υπάρχουν και αφιβολίες που λένε πως δεν γίνονται αυτό γιατί κάποια χώρα δεν θέλει ε, να επιτρέψει να είναι κάποιος πάνω από τους δικούς της εθνικούς συντονιστές. Να δούμε τώρα πώς θα βρεθεί η λύση. Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Και ένα μέτρο μπορεί να είναι να πούμε στα εθνικά one-stop shop πώς θα πρέπει να συνεργαστείτε καλύτερα για να επιτύχουμε αυτό τον στόχο της μεταφοράς των αγαθών καλύτερα από ότι τώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μαρινέσκου και όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί του για το δύσκολο αυτό θέμα εξίσου δύσκολο με όλα τα άλλα θέματα του σιδηροδρομικού πακέτου. Αν δεν καταφέρουμε να επιτύχουμε το One Stop Shop, την ενιαία θηρίδα, που είναι κάποια φιλοδοξία που ξεπερνάει την ευρωπαϊκή διαχείριση των διαδρόμων, αυτή η πρόταση για ενιαία θηρίδα αναδιάδρομο, για διαχείριση αναδιάδρομο, που ξεπερνάει το εθνικό επίπεδο, Μακάρι να γίνει και σε ορισμένους τομείς μια τέτοια πρόταση λειτουργήσε και σε άλλους όχι. Πάντως σίγουρα χρειαζόμαστε κάτι υπερεθνικό. Μια υπερεθνική πρόταση. Κύριε Μαρινέσκου, Κατέθεσα δύο τροπολογίε που πήραν αρνητικό πρόσημο, άρα διαφωνεί ο κύριο Μαρινέσκου, έτσι φαίνεται από τον κατάλογο ψηφοφορία. Ναι και θα αναθεωρήσετε όμω τη θέση σα για ορισμένε τροπολογίε, μήπως θα μπορούσατε να κοιτάξετε και τη δική μου. Στην 116, Απλώ στο τέλο προσθέτω κάτι που στο άρθρο 3 δεν το διευκρινίσατε δεόντω. δηλαδή λέω ότι ο διάδρομο θα πρέπει να, περιλαμ... να εντάσσεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα, στα σχέδια προτεραιότητα. Και επίση λέω ότι τα σχέδια προτεραιότητα ε, που λειτουργούν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων θα πρέπει να τροποποιηθούν για να προσαρμοστούν στους ε, σιδηροδρομικούς διαδρόμους. Αυτό ουσιαστικά λέω δηλαδή ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τα σχέδια και προγράμματα προτεραιότητας που θα καλύπτουν τα εμπορεύματα θα πρέπει να προσαρμοστούν στα χαρακτηριστικά του σιδηροδρομικού διαδρόμου, που είναι αυτονόητο. Και στην 158 τροπολογία θα ήθελα και τις ε, πολυλειτουργικές ε, πλατφόρμες να συμπεριλάβουμε υπόψη, εκτός από τους θερματικούς σταθμούς. Γιατί και εκεί λαμβάνεται υπόψη η επιβίβαση ή μάλλον φόρτο εκφόρτωση και από άλλους τρόπους μεταφοράς. Αυτές λοιπόν οι πολυ... ή μάλλον οι πολυδιαλειτουργικές πλατφόρμες ε, να εγκριθούν με την τροπολογία 158. Κύριε Κράμερ. Ξέχασα δύο πράγματα Συμφωνήσαμε σήμερα το πρωί στο άρθρο 13 παράγραφη 1 έως 5 να αντικατασταθεί το recognizing με το respecting. Αυτά συμφωνήσαμε με τον εισηγητή. Και στην συμβαστική λύση H, εκεί που μιλάει για να ληφθούν υπόψη τα silent freight trains. Και τέλος, ο κύριος Χαντραούι έχει δίκιο. Ε, όσο είναι τόσο άδικες οι συνθήκες πλαίσιο, όσο υπάρχει φορολογική προτίμηση για τους άλλους τρόπους, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον δίκαιος, ε, δίκαιη μεταχείριση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ευχαριστώ. Σύντομα και από μένα δύο σχόλια. Συμφωνώ με αυτούς που συνεχάρισαν τον ε, εισηγητή και τους σκιώδες εισηγητές και προσπάθειές τους. Μα ανησυχεί το θέμα τη οικονομική μεταφορά εμπορευμάτων στην Ευρώπη και αν υπάρχει μέλλον στην Ευρώπη. Και όσο λιγότερη δράση προωθήσουμε, τόσο λιγότερο, ε, λιγότερες πιθανότητες έχει να επιβιώσει αυτός ο τρόπος σε 20 χρόνια. Όπως είπε ο κ. Λιμπεράτσκι, με ανησυχεί και εμένα το γεγονός ότι η προσπάθειά μας για να αναπτύξουμε τους σιδηροδρόμους ε, περιορίζεται ε, στους φορείς τους δρομικούς ε, περισσότερο ε, μόνο και στα κράτη-μέλη. Όπως υπόθηκε, είναι ένα μικρό βήμα προς τα, προς τα εμπρός. Εγώ θυμάμαι το μεγάλο βήμα του Νίλ Άμστρονγκ στο φεγγάρι. Ένα μικρό βήμα μπορεί να αποδειχθεί γιγαντιαίο βήμα για την ανθρωπότητα. Ε, η Κομισιόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέσκο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους σκιώδεις εισηγητές και όλη την Επιτροπή Μεταφορών, γιατί μετά την πρώτη ανάγνωση, ο τρόπος που εξελίχθηκε ε, η δεύτερη ανάγνωση, που ξεκίνησε δύσκολα, μας ε, γεμίζει με ελπίδα, γιατί μπορεί να σημειωθεί πρόοδος. Θα έρθω και σε πιο συγκεκριμένες τροπολογίες, αλλά πιο γενικά θέλω να πω τώρα ότι η συζήτηση για αυτή την πρόταση καονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά το θέμα του αν θα διατηρήσουμε το status quo στον ε, συνδεδομικό τομέα ή όχι. Δηλαδή, οι ρυθμιστές των ε, υποδομών και οι συνδεδομικές εταιρείες ε, λειτουργούν σε εθνική βάση και δευτερευόντως σε ευρωπαϊκή βάση. Εάν θα οργανώσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις μεταφορές μέσω συντονισμού και εργαλείων συντονισμού και ρυθμιστικών, αν χρειαστεί, μέσων. Η Επιτροπή Μεταφορών ήταν πολύ επικριτική στην τελευταία συνεδρίαση για την εφαρμογή που θεωρώ ότι δεν είναι ικανοποιητική σε ό,τι αφορά το πρώτο πακέτο για τους ιδιοδρόμους. Τώρα έχει την ευκαιρία λοιπόν να βοηθήσει, να κινηθούν τα πράγματα για να εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία και να ανοίξει η αγορά στους σιδηροδρόμους. Να υπάρξει ανταγωνισμός να υπάρξουν διεθνείς ε, μεταφορές δεχόμενοι αυτή την έκθεση και τις τροπολογίες που προωθούν αυτή τη λογική. Υπάρχουν δυστυχώς όμως ε, τροπολογίες προς την αντίθετη κατεύθυνση και θα έπρεπε κατά την άποψη της Κομισιόν να τις προσέξουμε λιγάκι αυτές τις τροπολογίες. Θα τις αναφέρω αυτές τις τροπολογίες. Πολύ σύντομα για το One Stop Shop, την ενιαία θηρίδα. Να υπενθυμίσω ότι η αρχική πρόταση της Κομισιόν η οποία δεν έγινε δεκτή στην κοινή θέση του Συμβουλίου ήταν να έχουμε πραγματικά ένα one-stop shop, μία ενιαία θηρίδα, διάδρομο. Ούτω ώστε αυτό ο οργανισμό να έχει και δυνατότητα λήψη απόφαση για τη διαχείριση τη ε, κυκλοφορία από την αρχή στο τέλο του διαδρόμου. Σήμερα έχουμε τέτοιε θηρίδε, εθνικέ όμω, οι οποίε ασχολούνται με διάφορου διαδρόμου. Αλλά σε εθνικό επίπεδο μόνο. Αλλά δεν λειτουργούν, δεν λειτουργούν καθόλου αυτοί, αυτές οι θηρίδες που υπάρχουν χρησιμοποιούνται μερικώς και κατακαιρματισμένα από τις θηρομικές εταιρείες που ζητούν κάποιες αποφάσεις και ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις για, αυτό, για αυτές τις ενιαίες θηρίδες επισύρει διάφορες κριτικές ό,τι αφορά την κράτηση δυναμικού υπέρ κάποιων επιχειρήσεων και εις βάρος κάποιων άλλων ε, ή γίνονται κρατήσει, ε, αλλά δεν χρησιμοποιούνται μετά από τις αερομικές εταιρείε κτλ. Ε, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να δίνονται, να χορηγείται δυναμικό με τρόπο διαφανή αναδιάδρομου. Αυτό το, λόγο θα πρέπει, αυτό το ρόλο μάλλον θα πρέπει να τον παίξουν οι θηρίδες και να ελέγχονται από τους ρυθμιστικές αρχές ούτω ώστε ε, να μην υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού. Υπάρχουν τροπολογίε, όπω αυτή οι 140 και 142 που θέλουν να αποκλείσουν την, ε, ε, τον έλεγχο των θηρίδων αυτών από τι ρυθμιστικέ αρχέ. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να περιφερθεί ο, ο τομέα, Ο εγκεκριμένο υποψήφιο. αυτή είναι μια έννοια πολύ σημαντική για την πρόταση. Αυτή τη στιγμή οι υποψήφοι σήμερα μπορεί να είναι operator που δεν είναι ισοδρομικέ εταιρείε όμω. Ε, που μπορούν να ζητήσουν όμως διαδρόμους για να τους για να του δώσουμε μετά σε μια σιδηροδρομική εταιρεία και λαμβάνουν την έγκρισή του σε εθνικό επίπεδο. Αλλά όχι κατά, κατά ε, κατά μήκο ενό διαδρόμου. Θα πρέπει οι ίδιε ε, προποθέσει ανταγωνισμού να ισχύουν σε όλο το διάδρομο, αν θέλουμε να, να λειτουργούν. Και να υπάρχουν αυτοί οι εγκεκριμένοι υποψήφοι που μπορούν να κινηθούν για όλο το διάδρομο. Αυτό είναι πολύ σημαντική πρόταση τη Κομισιόν και χαίρομαι που με στηρίζει η δική σα ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Θα επιμείνω και θα πιέσω το Συμβούλιο για να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό. Υπάρχουν κάποιε συμβαστικέ ιδέε που υπερίπτανται, αλλά θα πρέπει να πιέσουμε αν θέλουμε να υπερβούμε το status quo. Αν δώσουμε έκριση σε αυτού του υποψήφιους, του εγκεκριμένου, τι νόημα έχουν αυτοί οι εμπορευματικοί διάδρομοι, αυτό το όργανο διαχείρισης για μας θα πρέπει να είναι ένα δουσού. Μία αρχή διαχείρισης που θα έχει δυνατότητα λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει λοιπόν γι' αυτό να έχει ένα νομικό, μια νομική υπόσταση και δεν θα πρέπει να μπλέξουμε διαφορετικά συμφέροντα. Στο Managing Board δεν θέλουμε να μπαίνουν ισοδομικές εταιρείες γιατί αυτές είναι πελάτες του Δουσού και των διαχειριστών υποδομών. Θα πρέπει να είναι μακριά τους, ούτω ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Φυσικά οι ισοδομικές ε, επιχειρήσεις θα μπορούν να πούν και αυτές κάτι, γιατί είναι οι πελάτες των διαδρόμων. Αλλά μπορούμε σε συμβουλευτικά συμβούλια να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτές τις ε, ε, περιστρομικές εταιρείες να πούν και αυτές την άποψή του, χωρίς όμως να δημιουργούν πρόβλημα στον αλήθεια ανταγωνισμό. Ένα λεπτό θέμα τώρα, που προέκυψε από την πρώτη ανάγνωση και για το Συμβούλιο και για το Κοινοβούλιο. Είναι οι κανόνες προτεραιότητας. Ο συμβιβασμό ο οποίος, ε, στον οποίο κατέληξε το Συμβούλιο δεν ικανοποιεί αρκετά την Κομισιόν. Είναι πολύ ε, εύθραυστη αυτή η ισορροπία. Και το είπε και το αναγνωρίζει ο εισηγητή. Και όμως οι τροπολογίες, οι τροπολογίες του δεν απομακρύνονται πολύ από την κοινή θέση. Υπάρχουν όμως άλλες που είναι αρκετά επικίνδυνες. Δεν θέλουμε να πούμε τώρα με αυτό ότι οι εμπορευματικές, οι μεταφορές θα πρέπει να έχουν την προτεραιότητα εναντί των μεταφορών επιβατών. Αυτό είναι αδιανόητο. Απλώς λέμε ότι κατά μήκο του διαδρόμου οι διαχειριστές των υποδομών θα πρέπει να συμφωνήσουν για να υπάρχουν κοινοί κανόνες προτεραιότητας που δεν θα θέτουν συστηματικά σε δεύτερη μοίρα τα εμπορεύματα έναντι των ε, ε, επιβατών. Όχι προνόμια για τα εμπορεύματα, αλλά να μην τα ρίξουμε σε δεύτερη μοίρα. Γι' αυτό η τροπολογία 151, 153 που εξαιρούν ε, τους κανόνες προτεραιότητας της ώρες εχμής αποδυναμώνουν εντελώς τον κανονισμό και τον καθιστούν ανώφελο. Και είναι προβληματικές λοιπόν. Τώρα, για τις ρυθμιστικές αρχές. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή για όλο το συνδρομικό δίκτυο και φυσικά οι ρυθμιστικές αρχές συνδέονται με τα εθνικά δίκτυα. Χρειαζόμαστε ρυθμιστικές αρχές που συντονίζονται μεταξύ τους. Τελειώνω, Πρόεδρε. Βλέπω ότι αδειμονείτε, Πρόεδρε. Τελειώνω, τελειώνω. Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πολυάριθμε τροπολογίε για την χάραξη των διαδρόμων είναι πολύ σημαντικές προφανώς για τους ε, βουλευτές που τις παρουσίασαν, ε, αυτονόητο είναι, αλλά για μας η σημασία των, των διαδρόμων ε, δεν έγκυται στην γεωγραφική τους θέση, αλλά στην επιχειρηματική τους, στις επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούν και στις, στη ζήτηση της αγοράς. το θέμα δεν είναι να ικανοποιήσουμε τον Α ή τον Β, τον Α ή τον Β βουλευτή, ας πούμε, οποιονδήποτε. Καταλάβατε. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πασκαρέλη. Σε... Ε, προσπαθώ να τηρήσω το χρονοδιάγραμμα, κάτι που δεν συμβαίνει συνήθως ε, στην ακρίβεια με την οποία γίνονται τα δρομολόγια στις διάφορες μεταφορές, γι' αυτό με είδατε να κουνάω το σφύρι. Ο εισηγητής ο κύριος Μαρινέσκου. Ο κύριος Χαδράουι είπε ότι ξεκινήσαμε από την ιδέα της βελτίωσης της ε, προτέρας κατάστασης του Σάτου Κουβό και ε, αν γίνει κάποιο συντονισμός των επενδύσεων και βελτιωθούν τα προγράμματα μεταφορών και αν σκεφτούμε και τη δυνατότητα της ύπερξενιας θηρίδας, του One Stop Shop και μόνο αυτά συνιστούν πρόοδο και μόνο αυτά βελτιώνουν την προτέρα κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε κάποιε επιφυλάξει και ανησυχίε που ελπίζω ότι θα διασκεδαστούν στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ όλους θερμά για τα σχόλιά σα και ευχαριστώ και πάλι του και οδησίγητες. Ευχαριστούμε κύριε Μαρινέσκου. Να σα υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία του σημείου αυτού θα γίνει αύριο στις 9 θα είναι η πρώτη ψηφοφορία. Οπότε μην ξεχάσετε και τις ηλεκτρονικές σας κάρτες ψηφοφορίες γιατί μπορεί να είναι πιο επίπονη ψηφοφορία και να διαρκέσει πιο πολύ από ό,τι είμαστε συνηθισμένοι συνήθω στι ψηφοφορίε. Γι' αυτό εννέα ραντεβού αύριο το πρωί μαζί με τι ηλεκτρονικέ σα κάρτε ψηφοφορία. Επόμενο σημείο, το σημείο 5, το βιώσιμο μέλλον για τι μεταφορέ. Ο κύριο Γκρό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με τη γραμματεία είχαμε πει να γίνει σήμερα μια συζήτηση μετά στις επόμενες 14 ημέρες ε, θα συζητήσω εγώ τις συμβαστικές προτάσεις με τους συναδέλφους. Μετά τον Ιούνιο λέμε να ψηφίσουμε. Με συγχωρείτε κύριε Γκρός, λέει ο πρόεδρος, εάν θέλετε να συζητήσετε σας παρακαλώ έξω από την αίθουσα. Όπως συχνά σας υπενθυμίζω, εδώ μέσα γίνεται μόνο μία συνεδρίαση, μόνο μία συνάντηση, συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Οτιδήποτε άλλο εκτός. Οπότε μετά λέει ο κύριος να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Ιουλίου και ελπίζω να τα καταφέρουμε. 376 τροπολογίες. Τέλος πάντων, ας μην είμαστε πολύ απεσιόδοξοι γιατί νομίζω πως πολλές από αυτές πήγαινουν προς παρόμοια κατεύθυνση π.χ. δεκάδες έχει μόνο η παράγραφος 20 που ορίζει τους στόχους. Οπότε νομίζω πως εκεί πέρα θα μπορέσουμε να βρούμε ε, μια συμβαστική λύση. 142 είναι αυτές που έχουν νέες ιδέες και άλλα είναι διάφορα γλωσσικά. Όσον αφορά τις νέες προτάσεις είναι σαφές για εμένα πως ε, ε, μιλάμε εδώ πέρα για την παραπομπή στη στρατηγική 2020 που πρέπει να γίνει για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Νομίζω πως ε, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για να εργαζόμαστε όλοι με τα ίδια νούμερα. Για να φύγουν εδώ πέρα τουλάχιστον ε, αρκετές τροπολογίες. Πράγματι και εδώ πέρα οι συνάδελφοι ενδιαφέρονται και για τα κοινωνικά. Αυτό παίζει ρόλο και για την ανάπτυξη πέθρου και για τις πτυχές της αστικές. Ολοκλήρωση τώρα της αγοράς δεν πρέπει να το αφήσουμε και αυτό το θέμα εξακολουθεί να παραμένει σημαντικός στόχος για εμάς αλλά δεν είναι ο μοναδικός ε, στόχος. Παράλληλα νομίζω μπορούμε να πούμε πως κινείται η ολοκλήρωση της αγοράς με κάποιες βελτιώσεις στο περιβάλλον, στα κοινωνικά και στον ε, ε, τομέα των τελών, εάν βεβαίως ε, μπορέσουμε να καταλήξουμε. Οπότε εκεί καθώς θα υπάρξει μάλλον μια ισοπερίκευση του εξωτερικού κόστους και δεν το βλέπω πάρα πολύ εύκολο αυτό, ειδικά με την προβληματική του διοξιδίου του άνθρακα, με τα θέματα της ασφάλειας, όλα αυτά που έχουν απόλυτη προτεραιότητα. Οπότε μάλλον για το θέμα της ασφάλειας θα έχουμε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο και εκεί πέρα θα πάνε όλες οι σχετικές τροπολογίες. Επίσης θα μπορούσε εδώ πέρα να αναφερθεί ένα νέο πρόγραμμα ή ένα δεύτερο πρόγραμμα για την οδική ε, ασφάλεια στους στόχους. Επίσης ε, αναφέρουμε τους πράσινους διαδρόμους, πρέπει οπωσδήποτε και αυτοί εδώ πέρα να βρουν μια θέση όπως και οι άλλες πτυχές όπου όμως λέμε πως πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ του σημαντικού και της πολύ μεγάλης λεπτομέρειας για αυτή την ε, χρονική στιγμή. Καθώς θα δούμε νομίζω ούτως ή άλλως τη Λευκή Βίβλο και εκεί πέρα θα μπούμε σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Κάποια άλλα σημεία σημαντικά θέλω να τα αναφέρω είναι οι οικονομικές αυτές πτυχές γιατί ανεξαρτήτως από τις μελλοντικέ εκτελήξεις θα πρέπει να δούμε ποια είναι η χρηματοδότηση να υπενθυμίσω πως ε, το ταμείο αυτό δεν είναι ένα τελείως νέο μέσο μπορεί να είναι ε, και επίσης εδώ πέρα να συμφωνήσει η Κομισιόν μπορεί να συσταθεί από τα υπάρχοντα μέσα των μεταφορών. Πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί με τα μέσα της ε, περιφερειακής πολιτικής, της συνοχής. Πρέπει να δημιουργηθεί εκεί πέρα μια γέφυρα και ελπίζω να υπάρξει μια προσθέμενη αξία και στα δύο επίπεδα. Οπότε θα το ξαναδούμε αυτό. Ειδικά επίσης ε, τα νέα μέσα, εγγυήσει και το τι θα γίνει και με τους επιβάτες αλλά και με τους κινδύνους της πρώτης φάσης πάρα πολλών έργων. Ένα άλλο θέμα είναι η λεγόμενη ε, αποτελεσματική συντροπικότητα, εάν θέλετε, όπως το λέμε αυτό. Δηλαδή πρέπει να δούμε εδώ πέρα πώς εξαρτώμαστε από όλους τους τρόπους ε, μεταφορών και όλοι τρόποι μεταφορών και ειδικά οι οδικές πρέπει να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον και να τονιστεί βεβαίως η πτυχή της ασφάλειας και να ε, βοηθηθεί οπωσδήποτε περισσότερο. Είμαι επεπισμένος δε πως ε, θα υπάρξει μία αλυσίδα εφοδιασμού των πόλεων και με αγαθά και στην μεταφορά προσώπων και αυτά μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά μέσα για την αποτελεσματική αυτή συντροπικότητα και υπάρχουν και τα περιβαλλοντικά κριτήρια, υπάρχουν και τα κοινωνικά κριτήρια που πρέπει να γίνουν σεβαστά. Οπότε να δούμε αυτό το οποίο είχαμε πει και στο παρελθόν, η οικονομία φαινός, από την άλλη βεβαίως και η φορολογία και το περιβάλλον και προτελευταίο σημείο μετά οι μετρήσιμοι στόχοι τους ανέφερα. Νομίζω πως πρέπει να δούμε ούτως ή άλλως νομίζω όλες οι ομάδες με τις οποίες ήρθα σε επαφή επί της αρχής συμφωνούν. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους σκιώδους συζητητές για τις πρώτες συναντήσεις που είχαμε. Ε, οι στόχοι εδώ πέρα που ορίζονται είναι σημαντικό θετικό σημείο παρά το ότι βεβαίω γνωρίζουμε πως είναι επικίνδυνο πάντα να ορίζει κανείς τους στόχους στην πολιτική αλλά πρέπει εδώ πέρα να τους ε, ορίσουμε κάπου. Τέλος ε, έχουμε αυτή την περίφημη υπηρεσία. Εγώ δεν θέλω να δημιουργηθεί μια άλλη ε, νέα υπηρεσία. Δεν θέλω. Επί της αρχής είμαι κατά αλλά στον τομέα των οδοικών και άλλων μεταφορών θα πρέπει σιγά σιγά οι ανεξάρτητες αυτές αρχές να γίνουν ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή. Ξέρω πως δεν αρέσει σε κάποιους να το ακούνε αυτό, αλλά γίνονται οι προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά αποτυχάνουμε γιατί η εθνική ερμηνεία ή τα εθνικά αντανακλαστικά αν θέλετε είναι κάπως πιο προστατευτικά. Αυτή είναι νομίζω η πέμπτουσία και η αποτελεσματικότητα της δουλειά μας εδώ πέρα. Εν ολίγης. Εάν έχουμε αύριο μια υπηρεσία που θα καταγράφει μόνο στατιστικά στοιχεία, δεν τη χρειαζόμαστε άμα είναι να βγάζει μόνο χαρτιά. Αλλά εάν έχουμε μια υπηρεσία η οποία θα ρυθμίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω μπορούμε να το σκεφτούμε και νομίζω πως ε, συμβαστική λύση μπορεί να πάει και προς την ε, κατεύθυνση την οποία θέλουμε για την Ευρώπη 2020. Πρέπει να δούμε βέβαια και την ουσία κάποια στιγμή το περιεχόμενο. Λοιπόν, αναμένω τις επόμενες 14 ημέρες ε, αυτά τα οποία θα μου πούν οι συζητητές, να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να συζητήσουμε συμβαστικές τροπολογίες και με αυτό τον τρόπο νομίζω θα μπορέσουμε να έχουμε και μια πολύ πιο μικρή, ένα πολύ πιο μικρό κατάλογο ψηφοφορίας από αυτό το οποίο φοβάμαι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γκρός. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειές σας να συντομεύσετε κάπως τον εκτενέστατο κατάλογο ψηφοφορίας. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Άλβαρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε τον κύριο Γκρός. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσπάθειά του να καταλήξει συμβαστικές λύσεις σε ένα κείμενο που αν είναι συνενετικό θα δώσει μεγαλύτερη ε, ισχύ στη θέση του Κοινοβουλίου και δυνατότητα επιρροή στο μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μεταφορές. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες που στόχο έχουν να συμπληρώσουν το κείμενο του κυρίου Γκρός και του είπα ότι θέλουμε να προσδιορίσουμε με σαφήνεια το στόχο και της ασφάλειας αλλά και το στόχο της εδαφικής συνοχής. Γιατί οι δύο στόχοι είναι συμβατοί μεταξύ τους και συνάδουν και με την αηφορία στις μεταφορές, με το βιώσιμο μέλλον τους. Υπό το ευρωπαϊκό πρίσμα φυσικά και υπό το πρίσμα των μεταφορών. Ο κύριος Γκρός μίλησε για μια καινοτομία, το χρηματοπιστωτικό ταμείο. Όταν ε, προσδιορίζεται μια πολιτική, εφοδιάζεται και με το απαραίτητο χρηματοπιστωτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο χρειαζόμαστε ένα ιδιαικό ταμείο, αλλά θα πρέπει να προσδιορίσουμε και ένα συγκεκριμένο ποσοστό που να το εγγυηθούμε κιόλα, γιατί είναι χαλεπή η κυρία από οικονομική άποψη. Οπότε καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη το golden rule. Είναι πολύ χρήσιμο για να έχουμε και μια ποιοτική διάσταση ε, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στις ε, υποδομές των μεταφορών που η απόσβεσή τους είναι μακροχρόνια και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις ε, επενδύσεις ως συνηθισμένες δαπάνες στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Κάτι άλλο που δεν αποσαφηνίζεται στην έκθεση είναι αυτό το θέμα της αποτελεσματικής διαλειτουργικότητας και των συνδυασμένων μεταφορών. Τι ακριβώς εννοείται με τις αποτελεσματικές συνδυασμένες μεταφορές, γιατί στόχος είναι να επιδιώξουμε μία ισορροπία μεταξύ των μέσων μεταφοράς, υποστηρίζοντας ιδιαίτερα τις ναυτιλιακές μεταφορές και τις ιδιοδρομικές μεταφορές. Γιατί αυτές οι δύο μεταφορές είναι ο καλύτερος τρόπος για να υλοποιήσουμε το στόχο, το στόχο μας για συνδυασμένες μεταφορές. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, των επιβατών και φυσικά να στηρίξουμε τις ε, δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτά νομίζω θα είναι τα κέρια σημεία και στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Φυσικά, ο η ε, κατάλληλη στιγμή, ο κατάλληλος χρονισμός είναι πολύ σημαντικό στην πολιτική και στην κατάλληλη στιγμή πέφτει η κυρία Γκρίσμπαχ από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πολύ σύντομα. Ε, ζητώ συγγνώμη. Καθέσα λιγάκι γιατί σήμερα έχει μεγάλη κυκλοφοριακή ε, συμφόρηση. Οι σημερινές μεταφορές, έτσι δεν μιλάω καν για τις μελλοντικές. Ε, Μπαίνω λοιπόν από τα μισά της συζήτησης. Ε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Ματιό Εγκρός για την ε, θαυμάσια δουλειά του και να υπενθυμίσω ότι κατά την άποψή μας και κατά την άποψη της ε, πολιτικής μου ομάδας των φιλελεύθερων που είμαι σκιώδης εισηγητής του, θέλω να πω ότι είναι στρατηγικά σημαντικό το να έχουμε μεγάλη ευρεία πλειοψηφία για αυτή την έκθεση που έχει μεγάλη σημασία και μακροπρόθεσμα, ούτως ώστε να έχουμε δυναμική θέση για αυτό το φάκελο. Ε, φάκελος που είναι πάρα πολύ στρατηγικός. Ο Μάτιο Γκρός ε, υπενθύμισε ότι υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες. Συμφωνώ με αυτό που ζήτησε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες και για να είμαστε και πιο δυνατοί αλλά και πιο ευανάγνωστοι και για να διατηρήσουμε όσο μπορούμε την έκθεσή μας ε, σε λίγες σελίδες που μιλάει για την ιστορία των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται να έχουμε ένα είδος χριστουγεννιάτικου δέντρου που θα αρέσει σε όλους. Να προσπαθήσουμε να ενωθούμε για να είμαστε συνεκτικοί, λακωνικοί και ή δυνατόν να προσδιορίσουμε με μεγάλη ενάργεια τις προτεραιότητές μας. Αυτά για τη μορφή και τη στρατηγική. Τώρα ας μπω στην ουσία. Με δύο λόγια. Ίσως ε, το είπαν και άλλοι βέβαια. Η ομάδα μου είναι ικανοποιημένη με τον βασικό στόχο. Δηλαδή να θεωρηθεί ότι είναι εκ των όνου κάνευ το να ληφθεί υπόψη η κλιματική αλλαγή στην πολιτική μεταφορών και να μειώσουμε το, το διοξίδιο του άνθρακα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Ίσως να βάλουμε και κάποιους ενδιάμεσους στόχους όμως. Ίσως αυτό το επιτύχουμε μέσω της συζήτησης που θα κάνουμε για τις τροπολογίες εφόσον καταλήξουν. Τώρα, εγώ προσωπικά θα ήθελα να τονίσω στην ε, σημασία του ευρωπαϊκού, ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, στον οποίο προστίθεται και το ευρωπαϊκό ε, δίκτυο. Ίσως ακόμη Γλάφ κανείς Αθήνας, αλλά η κρίση που γνωρίσαμε πριν από λίγες μέρες με το ηφαιστειακό σύννεφο έδειξε και, την, και το ευάλωτο αλλά και την αλληλεξάρτηση των κοινωνιών μας. Φυσικά, όταν ψάξαμε να βρούμε από τράγους, τράγους, ε, βρήκαμε την Ευρώπη, η οποία είπαμε ότι δεν συντώνησε αρκετά πράγματα, ενώ δεν είχαμε καμία τέτοια αρμοδιότητα. Ε, όταν μπορούμε λοιπόν, καλό είναι να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό συντονισμό. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς ε, επ' ευκαιρία των θεωρήσεων είχα υπενθυμίσει ο, πόσο σημαντικός είναι ο ευρωπαϊκός, ενιαίος ευρωπαϊκός ε, ουρανός. Άλλα σημαντικά σημεία τώρα. Φυσικά η ομάδα μου θέλει να προωθηθούν οι ολοκληρωμένες και πολύτροπες μεταφορές. Και θα ήθελα να βάλουμε τις αστικές μεταφορές σε πολλές ε, τροπολογίες. Να μιλήσουμε για την ασφάλειά τους και να φανταστούμε. Ε, ζητώ συγγνώμη, με κόβετε κύριε Πρόεδρε, δεν είχα καταλάβει ότι είχα τόσο λίγο χρόνο μόνο. Εντάξει, να μιλήσω τότε πιο γρήγορα. Αλλά βέβαια είναι επικίνδυνο για τους διερμηνείς. Θα τους κουράσω. Τελειώνω, Πρόεδρε. Να συμπεριλάβουμε όλα, όλες τις τεχνολογικές προόδους, ε, το καθαρό, καινοτόμο, πράσινο αυτοκίνητο και ή δυνατόν ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Ή δυνατόν. Για να λάβουμε υπόψη μας αυτό που είχε πει ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ή δυνατόν ένα σύστημα κυρώσεων σε όσους κάνουν διασυνοριακές παραβάσεις. Ούτω ώστε να αποκτήσει σάρκα και οστά αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα. Αυτές είναι οι προκαταρτικές παρατηρήσεις μου. Ε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης ε, θα επανέλθω ενδεχομένω, γιατί μπορώ να έχω και άλλα πράγματα να πω. Ευχαριστώ κυρία Λίχτεμπεργκερ για τους πράσινους. Ναι, ευχαριστώ πολύ την, ε, τον εισηγητή. Έκανε πολλά πράγματα για να βρούμε έτσι, κοινά σημεία. Εγώ τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στα σημαντικά για εμένα, καθώς πιστεύω πως πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε κάποια συνένεση. Εκεί στον συνολικό το τομέα της συντροπικότητας είναι υποχρέωσή μας ε, να αναφέρουμε τα μέσα μεταφοράς. Όλο σε ένα Eurospeak εκεί πέρα κινόμαστε και δεν το καταλαβαίνει κανένας πολίτης σε μια ευρωπαϊκή έτσι αργό. Να αναφέρουμε συγκεκριμένα τι εννοούμε. Να ξεκαθαρίσουμε. Με τα πόδια να πηγαίνει ο πολίτης. Και με το ποδήλατο. Αυτό σημαίνει συντροπικότητα και όχι μόνο ότι έχει ρόδες ή φτερά ή ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, τώρα πτερίγια δεν ξέρω κυρία συνάδελφε. Ε, άλλο που μου φαίνεται εμένα σημαντικό η αστική κινητικότητα για πόλεις άνω των 100.000 βεβαίω. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον ενημερωτικό σημείωμα που πρέπει νομίζω να μας απασχολήσει, να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Γνωρίζω πως πολλές πόλεις έχουν κάποιες προδιαγραφές, αλλά περιμένουν, ξέρω εγώ, 10-15 χρόνια και μετά βλέπουμε, θα κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Οπότε πρέπει να υπάρξει κάποια επιτάχυνση στην υλοποίηση αυτών των σχεδίων. Και αυτό θα γίνει αν στείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Τώρα τα μιλάμε για τα μέτρα. Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην συντροπικότητα, πάλι εδώ πέρα ευρωπαϊκή αργό, να πούμε ξεκάθαρα. Αποφυγή των μεταφορών ή μετατόπιση σε άλλα μέσα και βελτίωση. Και να πάμε σε ένα έτσι, ε, πακέτο συνολικό. Η συντροπικότητα από μόνη της ε, είναι μια ωραία λέξη. Αλλά όπως είπαμε, εγώ το Σαββατοκύριακο είχα κάποιες ε, συζητήσεις με πολίτες και πραγματικά ε, η διάλεκτος αυτή η ευρωπαϊκή τους ενοχλεί. Γιατί χάνονται στις λέξεις. Και μετά τα κράτη-μέλη κάνουν ό,τι θέλουν. Οπότε πρέπει να είμαστε πιο σαφείς διατυπώσεις μας. Και όχι μόνο η διατύπωση βεβαίω, ε, να αποφε... και τη ουσία να αποφευχθούν οι μετακινήσεις, να αποφευχθούν οι μετακινήσεις και μετά να δούμε τα υπόλοιπα. Γιατί υπάρχει καταναγκαστική ε, μετακίνηση. Να σας αναφέρω πώς έχει αλλάξει, αδειάσει, με το κέντρο των πόλεων και δημιουργούνται γύρω-γύρω προάστια και αναγκαστικά έχουμε μεταφορές. Για το Ταμείο τώρα των Μεταφορών. Το βασικό είναι να υπάρχουν σαφή κριτηρία εφορίας που θα αντικατοπτρίζονται και στη χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση δηλαδή για τους δρόμους να είναι σε ένα maximum 20 όπως έχουμε πει και τουλάχιστον μετά 15% για ποδήλατο και για τα πόδια. Να πάει σε αυτή την υποδομή. γιατί χάνονται εδώ πέρα αυτά τα πράγματα στα λόγια αυτά τα γενικά. Σας υπενθυμίζω εδώ πέρα τις τροπολογίες μας 320 και 334 που εμάς, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικές όσον αφορά τα όρια εκπομπών για να αυξηθεί, ε, να διπλασιαστεί νομίζω το ποσοστό υπεύθυνων οικολογικά μέσων μεταφοράς. Αυτό το οποίο επίσης είναι σημαντικό για εμένα όταν μιλάμε για το Ταμείο είναι πως η χρηματοδότηση σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μειωθεί τώρα επειδή έχουμε κρίση. Γιατί το, έχει εδώ πέρα μεγάλη μείωση. Πρέπει να παραμείνει ίδιο το ποσό αυτό το οποίο δίναμε τα τελευταία χρόνια. Νομίζω πως σε πάρα πολλά σημεία τα οποία συζητάμε εδώ πέρα μας έχουν επιβεβαιώσει αυτά τα οποία λέει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος στην ενδιάμεση έκθεσή της και απέτησή μας πρέπει να είναι να δούμε τους στόχους της μείωσης της αηφορίας για να τα πάρουμε σοβαρά αυτά και τη μείωση των εκπομπών. Και έτσι θα έχουμε μια πολύ ωραία έκθεση. Thank you. Mr. Ευχαριστώ κύριος Δεγκράντες Πασκουάλ. Ευχαριστώ. Ειλικρινά κύριε Γκρός, θερμά συγχαρητήρια. Και δεν το κάνω αυτό ούτε από αυρότητα, ούτε μόνο για να το κάνω για το πρωτόκολλο. Είναι πολύ σωστή η έκθεσή του, πολύ μεστή και προβαίνει σε μια ειλικρινή και επικριτική διάγνωση της κατάστασης ε, δίνοντας σαδρές γραμμές για τη λευκή βίβλο των μεταφορών για τα επόμενα δέκα χρόνια. ο εισηγητής ε, παρουσιάζει τη δική του θέση, που δεν είναι καθόλου βολονταριστική, επικεντρώνει την προσοχή στα κακό κείμενα και δίνει και κάποιες προτάσεις για τις βελτιώσεις και τις λύσεις. Και αναφέρεται στην ανάγκη ενός χρηματοπιστωτικού ταμείου. Υπάρχει πρόσκληση της αυξανόμενης ζήτησης των εμπορευματικών μεταφορών. Η λύση των συντροπικών μεταφορών που θα δίνει και για τα εμπορεύματα για τους επιβάτες λύση. Ανάγκη ασφαλών ζώνων ανάπαυλας. Μία διάγνωση που θα πρέπει να είναι οξυδερκής και να καταλήγει σε αλληλοσυμπληρούμενες μεταφορές και τρόπους μεταφοράς. Επίσης θα πρέπει να βρεθούν κάποια, να βρεθούν κάποια κριτήρια αποτελεσματικότητας Πολύ σωστή είναι και η διαπίστωση ότι δεν είναι πάντα οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι ναυτιλιακές μεταφορές που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και είναι πολύ πιο φιλοπεριβαλλοντικές από τις οδικές μεταφορές. Κάτι που δεν είναι κρατούς άποψη. Επίσης, η αποτελεσματική συντροπικότητα θα πρέπει να είναι η έννοια του μέλλοντος και να μην στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, αλλά σε μια αλληλοσυμπλήρωση που θα χαρακτηρίζεται κυρίως από την ανάγκη αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι η συντροπικότητα για μένα ε, εννοούμε συμβίωση, μια αρμονική συνύπαρξη. Αυτό είναι το ζητούμενο όταν μιλούμε για αποτελεσματική συντροπικότητα. Ο κύριος Γκρός ε, ε, αναφέρει με επισημότητα ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ένα αποτελεσματικό δίκτυο υποδομών και για να βελτιώσει τις υπάρχουσες υποδομές θα πρέπει να αυξήσει τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις επενδύσεις στις υποδομές. Αυτό το αναφέρω και στις α, τροπολογίες μου, τις πέντε, που έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά ε, δεν έχω καμία αξίωση να γίνουν δεκτές α, πλήρως. Γιατί φυσικά ο κάθε ευρωβουλευτής εύλογα υπέβαλε τις τροπολογίες που έκρινε σκόπιμες. Και πολλές από αυτές ε, είναι πανομοιότυπες και αυτό που θα αναζητήσει ο εισηγητής είναι μια συνένεση, μια συμβαστική λύση ώστε να ικανοποιηθούμε όλοι όσοι έχουμε παρόμοιους στόχους. Και είπε ο κ. Γκρός ότι θα ανταποκριθεί στα αιτήματα και των σχεδόν εισηγητών και των ε, ε, συντακτών τροπολογιών. Πιστεύω ότι θα βρει ικανοποιητικού τρόπους ώστε όλοι να βρούμε ένα σωστό αντικατοπτρισμό σε αυτό το σχέδιο που θα αποτελέσει τη βάση για την επόμενη Λευκή Βίβλο. Εγώ περιορίζομαι στα πέντε σημεία που θίγω στις τροπολογίες μου. Δεν θα πρέπει να ε, βάλουμε σε δεύτερη μοίρα κανένα τρόπο μεταφοράς. Καμία Μία μέθοδος μεταφοράς να μην υποστεί διακριτική μεταχείριση. Αν δεν βρούμε αντικατάσταση, να μην ε, υπάρξει διάκριση αρνητική σε έναν τρόπο μεταφοράς. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμόσουμε πυγμή και να εφαρμόζουμε σωστούς ελέγχους. Για παράδειγμα, είχαμε τον ταχυγράφο. Θα πρέπει να βρούμε ελαστικούς τρόπους για να συμφιλιώσουμε την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή, κάτι που προηγουμένως δεν ήταν δυνατό. Επίσης, θέλουμε και ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο επενδύσεων με μια ενίσχυση των μέτρων που θα τάσσονται υπέρ της τεχνικής διαλειτουργικότητας. Τέλος, για την ε, επίτευξη αποτελεσματικών αυτιλιακών μεταφορών είναι απαραίτητο να απελευθερωθεί η διαχείριση των λιμένων. Επίσης είναι απαραίτητο να αυξήσουμε τους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς πόρους και να γεφυρώσουμε τα χάσματα που υπάρχουν μεταξύ μερικές φορές και όμορων περιεχών και ε, να κάνουμε τη σωστή διάγνωση της ανεπάρκειας των μέχρι τώρα πόρων. Το ηφαίστειο μας άνοιξε τα μάτια, κύριε Πρόεδρε, γιατί είδαμε δυστυχώς ότι είμαστε ανίκανοι μερικές φορές να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη στη μελλοντική συζήτηση. Ήταν ε, πολύ σημαντικό αυτό το πάθημα και θα πρέπει να μας γίνει μάθημα για να διορθώσουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστώ τον κύριο Γκρός γιατί μας υπέβαλε όλους σε σημαντικές πνευματικές ασκήσεις και νομίζω ότι κατάφερε να μας συμπαρασύρει όλους ε, με τις προτάσεις και τον ενθουσιασμό του και απόδειξη η πληθώρα των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί έχει αυτό το ταλέντο ο κύριος Γκρός να δίνει σημαντική τροφή για συζήτηση. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη χρηματοδότηση. Μιλήσατε για την ανάγκη ίδρυσης ειδικού ταμείου μεταφορών. Ήδη υπάρχει το ταμείο για τα δίκτυα. Αλλά εγώ άλλο εννοούσα, άλλο θα είχα εγώ στο μυαλό μου για ένα ταμείο μεταφορών για τις υποδομές στην Ευρώπη. Βέβαια, Ίσως θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό αυτό το ταμείο σε σχέση με τα περιφερειακά ταμεία. Έχουμε το Ταμείο συνοχή, όπου το 50% των κονδύλιων του χρηματοδοτεί υποδομές. Υπάρχει και το ΦΕΝΤΕΡ, το Αναπτυξιακό Ταμείο, που σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτεί και υποδομές. Βέβαια, σε ορισμένε περιπτώσεις όπως στη χώρα μου λειτουργήσαν καλά αυτέ οι επενδύσει, αλλά σε άλλε χώρε χρησιμοποιήθηκαν πολύ λιγότερο αυτέ οι δυνατότητε. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε συμπληρωματικό αυτό το ταμείο με τα περιφερειακά. Επίση, ε, με το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο, κατορθώσαμε ένα ποιοτικό άλμα και βρήκαμε και φρέσκο χρήμα. Γιατί υπάρχει με αναδιοργάνωση, υπάρχει ανακατανομή των κονδυλίων. Ίσως τώρα θα πρέπει να το εξετάσουμε για να φτάσουμε στο ένα και που είναι το ζητούμενο και που δεν το καταφέραμε στις προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικές για να χρηματοδοτήσουμε τις μεταφορές. Θα ήθελα να είμαστε πιο φιλόδοξοι και σε αυτό το Ταμείο των Μεταφορών να είμαστε ευρηματικοί, να δείξουμε φαντασία και τώρα που θα αναθεωρήσουμε τα δίκτυα να φροντίσουμε, να πείσουμε και το Συμβούλιο αλλά και τους συμπολίτες μας ότι θα πρέπει να μας βοηθήσουν. Για να τους πείσουμε όμως θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα υπάρξουν και νέα κονδύλια, γιατί τα περιφερειακά κονδύλια είναι περιορισμένα. Όσο και να τα τραβήξουμε, δεν μπορούν να, να καλύψουν τις ανάγκες μας. Θα πρέπει να τα εμπλουτίσουμε. Και χωρίς συμπλήρωση των κονδυλίων δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας. Οπότε θα πρέπει να προσθεριστούμε το Συμβούλιο σε αυτούς τους στόχους και να δείξουμε ευρηματικότητα και δημιουργικότητα. και να διευκολύνουμε με το Golden Rule και το Σύμφωνο Σταθερότητας. Αλλά δεν θα έχουμε μόνο το ευρωπαϊ... τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτή την προσπάθεια να πείσουμε λοιπόν το Συμβούλιο και τους συμπολίτε μας τι θέλει να κάνουμε. Ο κύριος Αλκαντράουι. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά του και για αυτή τη δουλειά που θα πρέπει να κάνει ακόμα να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Έχουμε πολλή δουλειά για να καταλήξουμε. Ποιο είναι το νόημα εδώ πέρα. Να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην Κομισιόν για το τι θέμε εμείς στα λευκή αυτή βίβλο. Προσωπικά θεωρώ πως μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ μεταφοράς προσώπων και εμπορευματικών μεταφορών. Ειδικά όσον αφορά τη μεταφορά προσώπων πρέπει να δώσουμε βάση στην ενίσχυση της ε, αστικής ε, κινητικότητας ε, που οπωσδήποτε την έχουμε συζητήσει να ενισχυθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι συντροπικές λύσεις και ήπιες μεταφορές, όπως π.χ. το ποδήλατο αυτό, πάντα σε συνδυασμό με δίκτυα υψηλής ταχύτητας για να μπορούν οι άνθρωποι να μετακινούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη με έναν ε, αηφόρο τρόπο όσον αφορά τα αγαθά. Αντιλαμβάνομαι πως ε, είστε υπέρ αυτής της αποτελεσματικής συντροπικότητας όπως λέτε, εντάξει τη στηρίζω, αλλά δεν ξέρω αν σημαίνει αυτό πως ε, θα πρέπει να υπάρξει αυτή η μετατόπιση προς αυτούς τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μεταφορών. Για να οδηγηθούμε σε ένα πιο αηφόρο σύστημα θα πρέπει να έχουμε ένα μείγμα μέτρων για την μείωση της ε, κατανάλωσης ενέργειας, να έχουμε έξυπνα συστήματα, ε, να ενσωματωθεί το εξωτερικό κόστος και βεβαίως επενδύσεις. Ε, αυτό μπορεί να γίνει η έξυπνη συντροπικότητα που λέτε μόνο εάν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των τρόπων μεταφοράς αλλά και ε, εντός των τρόπων που π.χ. τα γνωστά προβλήματα των σιδηροδρόμων που πρέπει να βελτιωθούν και βέβαια πρέπει να υπάρχει και χρηματοδότηση για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά εκεί πέρα είναι το, το κλειδί. Αυτή είναι η ουσία. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας, της εξασφάλισης, κοινωνικός διάλογος, τα δικαιώματα των επιβατών, κοινωνική συνοχή. Και τέλος νομίζω πως συμφωνούμε με το ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο στα καλά λόγια, αλλά να πάμε σε συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμους στόχους. Εγώ θα ήθελα η Κομισιόν να αναφέρει συγκεκριμένα πώς θα οδηγηθούμε στην επίτευξη αυτών των στόχων ε, και τι χρονοδιάγραμμα βλέπει η Κομισιόν. Γιατί το λάθος το οποίο κάναμε στην προηγούμενη λευκή βίβλο είναι πως είχαμε ένα ωραίο κείμενο, αλλά η αξιολόγηση μετά έδειξε πως πολλοί από αυτούς τους γενικούς στόχους δεν, δεν εφαρμόζονταν. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ασκήσουμε πίεση και ένας τέτοιος τρόπος είναι να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον κάθε στόχο. Οπότε αναμένουμε τώρα τις ερχόμενες εβδομάδες τις προτάσεις σας ε, για συμβαστικές ε, τροπολογίες για να μπορέσουμε μετά να δώσουμε συνέχεια. Και έχω μια έτσι πολύ καλή αίσθηση για αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Σίτα. Κύριε Μάισνερ, ευχαριστώ. Τέσσερα σημεία θέλω εγώ να αναφέρω. Πρώτον, ε, είπατε πως υπάρχουν 376 τροπολογίες. Ή έχει κάνει πολλά λάθη εδώ πέρα, ο συγγετής έχει ξεχάσει πολλά πράγματα. Α, δεν νομίζω, είναι πολύ καλή έκθεση. Είναι μια έκθεση που τη χρειαζόμαστε για το μέλλον των μεταφορών, έτσι, για, για να μην νομίζετε πως είναι όλα χάλια γνωρίζουμε πως ε, πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο μήκος οι εκθέσεις, οπότε κάποια πράγματα πρέπει να συμπληρωθούν μετά. Και μετά έχουμε πάρα πολλά λόγω του ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και βεβαίως η κινητικότητα για τους ανθρώπους και τα αγαθά είναι μια κατάκτηση την οποία πρέπει να διατηρήσουμε και στο μέλλον. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αποτελεσματική συντροπικότητα. Ακούγεται έτσι λίγο κάπως σαν Eurospeak που είπε και η συνάδελφος. Τι σημαίνει δηλαδή ακριβώς. Περιέχει αυτά τα οποία θέλουμε. Και την ασφάλεια και την κοινωνική διάσταση και την αηφορία. Οπότε πρέπει να το υποστηρίξουμε και κάτι άλλο που μου αρέσει ιδιαίτερα εδώ πέρα που μιλάτε για στην αποτελεσματική συντροπικότητα λέτε πως όλοι οι τρόποι μεταφορών είναι σημαντικοί και τους χρειαζόμαστε και αυτό παρατηρήσαμε και με την στάχτη. Π.χ. μπορεί κάπου εν μέρη να αντικατασταθούν τα αεροπλάνα από γρήγορα τρένα. Πράγματι, αλλά βλέπετε πως ε, ε υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορεί να γίνουν ε, π.χ. μόνο με άλλους τρόπους μεταφορών. Οπότε χρειάζονται πλατφόρμες ε, συντροπικές για να μπορεί να περάσει ο άνθρωπος από το ένα μέσο μεταφοράς στο άλλο. Γιατί ξέρουμε πως ε, λίγα πράγματα μπορούν να μεταφερθούν σιδηρόδρομους ε, ή στα πλοία γιατί δεν υπάρχουν δυνατότητες μεταφόρτωσης, με συγχωρείτε. Και για την συντροπικότητα εδώ πέρα που λέτε και εδώ πέρα η δική μου ομάδα είπε πως πρέπει να δούμε την δυνατότητα μεταφοράς στα πλοία και στην εσωτερική ναυσιπλοεία και αυτό το οποίο οπωσδήποτε θα ήθελα να υποστηρίξω είναι τα ποδήλατα στις πόλεις. Πράγματι μπορεί να γίνει αυτό στις ε, πόλεις, είμαι και ηλεκτρικό ποδήλατο. Και αυτή είναι μια πτυχή σημαντική για το μέλλον των μεταφορών. Σημείο 3. Η χρηματοδότηση. Αναφέρθηκε ένα ταμείο χρηματοδότηση. Το ανέφερε ο Σιμ Κάλλας όταν είπε πως πρέπει να επεκταθεί να επεκταθούν οι συγκοινωνίες και χρειάζονται ε, χρηματοδότηση. Ελπίζω εδώ πέρα πραγματικά να βρούμε κάποιες δυνατότητες. Χρειάζεται περισσότερα χρήματα ο κλάδος αυτός Πρέπει λοιπόν να βρούμε και ε, λύσεις ε, δημιουργικές. Και το τέταρτο σημείο που είναι για μένα εξαιρετικά σημαντικό είναι το πώς η εσωτερική αγορά θα ολοκληρωθεί στον τομέα των, ε, μεταφορά, μεταφορών. Δηλαδή μπορεί να έχει κανείς σε εθνικό επίπεδο ένα τέλειο ε, εθνικό σύστημα και μετά αλλάζει, αλλάζουν οι γραμμές στο των σιδηροδρόμων ή σταματάει στα σύνορα, πρέπει να κατέβει και να πάρει άλλο τρένο. Άμα δεν μπορεί να βγάλει ένα εισιτήριο από το βορρά μέχρι τον νότο, ο πιβάτης δεν έχει πάρα πολύ νόημα. Οπότε νομίζω είναι πάρα πολύ καλή η πρόταση του ε, εισηγητού και τον ευχαριστώ. Συμφωνώ και εγώ με τους ε, προλαλήσαντες ε, ότι ο κύριος Γκρός έκανε μια θαυμάσια προσπάθεια. Eh, και είναι πολύ σημαντική βάση για τη συζήτηση. Μιλάμε για, το, για τη Λευκή Βίβλο, για το βιώσιμο μέλλον των μεταφορών, για τις ε, Ανταγωνιστικέ εμπορευματικέ μεταφορέ, όλα αυτά τα θέματα που έχουμε επιτάπητο ε, είναι ανοιχτά ακόμα, τα συζητάμε. Αλλά το θέμα νομίζω είναι ένα τελικά. Γιατί ο ευρωπαϊκός χώρος είναι ένας και όλα τα επιχειρήματα που ακούσαμε ισχύουν για όλους τους τρόπους μεταφορών. Αυτό που λείπει είναι ένας εξορθολογισμός στον προγραμματισμό ούτω ώστε να πάμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κανένα πρόβλημα δεν έχω να τα συζητήσουμε όλα αυτά χωριστά. Αλλά τελικά θα πρέπει να υπάρξει μια συνισταμένη... Εδώ νομίζω ότι κάνουμε το αντίθετο. Ε, Ξεκινάμε από μια συζήτηση, ε, καταλήγουμε σε κάποιες συνιστώσεις και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στη συνισταμένη αυτή. Θα ήθελα να σας παροτρύνω όλους, όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα και για τον ανταγωνιστικό τρόπο των ε, μεταφορών των εμπορευμάτων και αυτό που μας μίλησαν, για το οποίο μας μίλησαν τις προάλλες, το μέλλον των μεταφορών TEN, όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη. Όταν μιλούσαμε προηγουμένως για την ανταγωνιστικότητα και την συντροπικότητα, αυτά είναι όροι κλειδιά, δεν χρειάζονται να τους εξηγήσουμε. Πρέπει να παντρέψουμε, να συνδέσουμε όλες αυτές τις ροές μεταφορών, ε, τα λιμάνια, τους αερολιμένες, ε, ακόμα να εντάξουμε μέσα αυτό το δίκτυο και το ποδήλατο, ας πούμε. Ε, θα πρέπει τις ροές αυτές και τους κόμβους να τους αλληλοσυνδέσουμε. Αν όμως αυτά τα δούμε χώρια, αλλιώς τις ροές, ε, τους επιβάτες αλλού, τη βιωσιμότητα κάποιων τρόπων διαφορετικά. Πώς μπορούμε να τα εντάξουμε όλα αυτά σε ένα συνεκτικό όλο. Γι' αυτό ακριβώ μίλησα για τον προγραμματισμό. Ε, για τη χρηματοδότηση τώρα. Με μεγάλη χαρά άκουσα τους ευρωβουλευτές στο Κοινοβούλιο ε, να μιλούν για αυτό το χρηματοδοτικό ταμείο. Έχουμε και ένα άλλο παράδειγμα ενό αντίστοιχου ταμείου του Μάργκεριτ. Τα χρήματα προέρχονται από τον προϋπολογισμό, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για να δούμε πώς μπορούμε ενδεχομένως ε, πέρα από τα χρήματα του προϋπολογισμού να συνδέσουμε, να μαζέψουμε χρήματα μέσα από τα ευρωομόλογα ε, και να τα χρησιμοποιήσουμε για αυτό το ταμείο. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα. Μιλήσαμε επίσης για το υβριδικό αυτοκίνητο, το, αυτοκίνητο, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο που καίει υδρογόνο. Μπορούμε και αυτά να τα δούμε να τα συζητήσουμε ως χωριστά επιχειρήματα, αλλά θα πρέπει να εντάξουμε στο βιώσιμο μέλλον των μεταφορών. Όλα αυτά λοιπόν πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε έτσι. Εγώ είμαι η συγγητής αυτής της έκθεσης ε, της Επιτροπής Ήτρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω την ασφάλεια, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις, ε, τη μείωση των ε, εκπομπών, την ενεργειακή κατανάλωση και κυρίως τις έξυπνες μεταφορές, τα έξυπνα συστήματα μεταφορών. Και αυτά να τα σας παρακαλώ υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τον Ματιό Γκρός για την οξυδέρκειά του, την ευφία του και την ενδιαφέρουσα πρότασή του. Όλοι βέβαια προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε την έκθεση αυτή και να εμβαθύνουμε. Και συμμερίζομαι την ευφυΐα με την οποία πολύ επισήμανα τον πολυδιάστατο χαρακτήρα. Αλλά το θέμα ήταν να ξαναφέρουμε τις μεταφορές στο επίκεντρο της Επιτροπής μας. Αν έκανα μια σωστή παρατήρηση με το μάτι του νέου εισερχόμενου, βλέπω ότι οι μεταφορές αρχίζουν και χάνουν κάπως την έγκλη τους. Και εδώ και γενικώ στα κοινωτικά θεσμικά όργανα. Το βλέπουμε και στην αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ουδέν σχόλιο. Αν δούμε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπιστώνουμε ότι χαλαρώνει το ενδιαφέρον της, αλλά και οι ουσιαστικές προτάσεις κλείπουν για πολλά θέματα που επισημάναμε. Οπότε, η έκθεση για το μέλλον των μεταφορών θα πρέπει να μεταφέρει το μήνυμα ότι δεν αρκεί να εξηγήσουμε ότι οι μεταφορές είναι μείζον ζήτημα και ότι είναι το 10% της οικονομίας, ότι συμβάλλουν στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της Ευρώπης, γιατί η κινητικότητα είναι και πολιτικό θέμα. Φυσικά είμαστε και ρηπαίνοντες, γιατί οι μεταφορέ αντιπροσωπεύουν το 27% της ρήπανση, αλλά δεν αρκούν αυτά να πούμε σε μια έκθεση για το μέλλον των μεταφορών. Σε μια έκθεση που αφορά το μέλλον των μεταφορών, το βιώσιμο μάλιστα μέλλον, και ο εισηγητή πολύ σωστά, αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες στη συζήτηση πολύ σωστά μίλησαν για τα οικονομικά. Γιατί αν δεν ακούγεται η φωνή μα σε πολιτικό επίπεδο, πολύ λιγότερο θα ακουστεί σε οικονομικό. Γιατί υπάρχουν προβλήματα και οικονομικά και δημοσιονομικά. Και αν δεν είμαστε πιστικοί σε πολιτικό επίπεδο, σίγουρα δεν θα βρούμε ούτε τα οικονομικά μέσα για να υλοποιήσουμε τους πολιτικούς μας στόχους. Αλλά αυτό είναι οριζόντιο πρόβλημα στα πολιτικά θεσμικά όργανα. Οπότε, πολύ σωστά όλα αυτά που είπατε για την έκθεση, αλλά υπάρχει και κάτι επιπλέον. Θα πρέπει να είναι ένας πολιτικός και οικονομικός φορέας για να, να διατρανώσουμε τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα, τους στόχους μας για το μέλλον της πολιτικής μεταφορών. Σας ευχαριστώ όλοι κύριε Τσικάου. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γκρός για την έκθεσή του και να σας παρουσιάσω εν συντομία τα σχόλιά μου θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τους δημοσιονομικούς μας πόρους και χαίρομαι που οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν και στο θέμα αυτό. Ο τομέας των μεταφορών θα πρέπει να αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών και γι' αυτό χρειαζόμαστε αντίστοιχα με τους φιλόδοξους στόχους μας κονδύλια για να τους υλοποιήσουμε. Ακόμη και αν οι επιπτώσεις της ηφαιστειακής τάχτης ε, δεν ήταν ε, τόσο ολέθριες από οικονομική άποψη, είχαν τεράστιο παρόλα αυτά αντίκτυπο στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, και στη μεταφορά εμπορευμάτων. 66% των ε, επιβατών που έμειναν εγκλωβισμένοι και μπλοκαρισμένοι στα αεροδρόμια έμειναν σε αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε συντροπικότητα. Γι' αυτό το 6% των ε, επιβατών που αποκλείστηκαν στα αεροδρόμια θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιήσει πιο ανεπτυγμένο σύστημα ε, σιδηροδρόμων ε, μεγάλης ταχύτητας και να φτάσουν στον προορισμό τους πολύ πιο εύκολα. Όταν μιλούμε για διαλειτουργικότητα ή συντροπικότητα θα πρέπει να αναζητήσουμε καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ των ναυτιλιακών μεταφορών και των μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών. Σε επίπεδο ναυτιλιακών μεταφορών έχουμε ευρωπαϊκή στρατηγική μέχρι το 2018, αλλά για τις εσωτερικές πλωτές οδούς για τις ποτάμιες μεταφορές, για παράδειγμα, δεν έχουμε αντίστοιχη ευρωπαϊκή στρατηγική. Οπότε είναι ενδιαφέρον, από την ευρωπαϊκή πολιτική, να αναζητήσουμε τους ακρογωνιαίους λίθους μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις μεταφορές ε, από τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και σε τρόπους πιο φιλοπεριβαλλοντικούς τρόπους μεταφοράς ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι αστικές συγκοινωνίες. Για παράδειγμα, γιατί να μην χρησιμοποιούμε περισσότερο τα ποδήλατα στις πόλεις για την μετακίνησή μας. Γιατί να μην επενδύσουμε και σε αυτό το τομέα. Ίσως χρειαζόμαστε και εκεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα ποδήλατα, για παράδειγμα. Όχι μόνο για τις αστικές μεταφορές, αλλά και για άλλου είδους συγκοινωνίες. Γιατί μας ενδιαφέρει ο πολιτιστικός τουρισμός, για παράδειγμα. Η ποδηλασία, και η Ισπανία είναι καλό παράδειγμα εδώ, είναι παράδοση. Και όταν κάποιος ε, σταθμεύει το αυτοκίνητό του, μπορεί δωρεάν να πάρει ένα ποδήλατο για να επισκεφθεί κάποια μνημεία που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, κάποια αξιοθέατα, είναι εύκολο να βρει χάρτη. Γιατί να μιμηθούμε αυτό το παράδειγμα και εμείς και να το αναπτύξουμε περισσότερο. Και τέλος, για την κινητικότητα στις πόλεις, πιστεύω ότι και εδώ χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όπου οι πολεοδόμοι και οι ρημοτόμοι θα πρέπει να συνεργαστούν με τους αρχιτέκτονες για να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και η σωστή πολεοδομία να παρακολουθήσει αυτές τις πολιτικές συγκοινωνιών. Κυρία Ευχαριστώ. Για αυτά που είπε ο κύριος Ρικέ, θέλω να ε, πω και εγώ κάποια πράγματα. Έχει δίκιο που λέει ότι αυτή η έκθεση θα πρέπει να γίνει ένα, να χρησιμεύσει ως εργαλείο. Και ευχαριστώ τον κύριο Γκρός για τη δουλειά του. Ε, θα προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες και να βρούμε συμβιβασμού. Αλλά θα πρέπει αυτή η δουλειά να θυμίζει την προσπάθεια που γίνεται για το 2020 για την ενέργεια. Ε, η Λευκή Βίβλος θα μας ε, ετοιμάσει τα επόμενα βήματα. Και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό. Μπορούμε να μιλήσουμε για ένα πακέτο κλίμα μεταφορές ε, και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτό το πακέτο με την έκθεση. Και ελπίζω με τις ε, τροπολογίες μας να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το καθεστώς της έκθεσης πρωτοβουλίας αλλά να καταστεί τελικά μία πολιτική στρατηγική, όχι τεχνική, έτσι. Ε, εντάξει, τώρα το περιεχόμενο συζητιέται. Αλλά το βασικό είναι να χρησιμοποιηθεί αυτή η έκθεση ως ε, μοχλός πίεσης. Η κυρία Γέγκερ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Εκ νέου, Πρόεδρε. Η Κομισιόν σημειώνει ότι με χαρά ότι 300 376 τροπολογίες που έγιναν για την έκθεση δείχνουν το ενδιαφέρον που υπάρχει και την τεράστια σημασία του θέματος. Καλωσορίζουμε τη θέση που εκφράζεται στο σχέδιο της έκθεσης που υποστηρίζει ούτως ή άλλως και, τον προσανατολισμό της Κομισιόν για τη στρατηγική του 2020. Η αύξηση της θα δημιουργήσει πίεση στο, στο δυναμικό. Αυτή η ζήτηση θα εξαρτηθεί από την, την αποτελεσματικότητα και την συντροπικότητα των μεταφορών. Κάτι που ακούστηκε. Η πίεση στο δυναμικό, στο, στο, στα δυναμικότητα των μεταφορών α, συνδέεται με τη συζήτηση για την επικουρικότητα, γιατί έχουμε περιορισμένες αρμοδιότητες. Ε, είναι πολύ σημαντικό ε, οι μεταφορές να γίνουν βιώσιμες ε, με διάφορους όρους, περιβαλλοντικούς, ασφάλειας κτλ. Και αυτό θα αντανακλάται και στην Λευκή Βίβλο και να έχουμε πιο ανταγωνιστικό σύστημα μεταφορών. Αυτό σημαίνει και ανοιχτές αγορές, όπως είπατε κι εσείς. Επίσης, σημειώνω διάφορες παρατηρήσεις σας τις διασυνοριακές παραβάσεις, αύξηση της ε, ε, χρηματοδότησης, ε, τεχνολογικές εξελίξεις. Συμφωνώ με αυτές. Και θα μας επηρεάσουν πάρα πολύ και η επιρροή του ηφαιστείου. Όπως υπόθηκε, δεν θέλετε να υπάρξει και άλλη μία agency, αλλά το πιο σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσουμε την επικουρικότητα. Σε ό,τι αφορά το δύσκολο θέμα της χρηματοδότησης ε, των υποδομών των μεταφορών, ε, όλοι συμφωνείτε ότι στα πλαίσια της ε, παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Επομένως, εκ μέρους της Κομισιόν το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οι στόχοι μας παραμένουν οι ίδιοι. Η Κομισιόν θα τονίσει το θέμα της χρηματοδότησης που τόνισε και ο αντιπρόεδρός μας. Αναγνωρίζοντας όμως τις δυσκολίες και το τι σημαίνει συνοχή, ειδικά για κάποια νέα μέλη. Ακριβώς γι' αυτό δεσμευόμαστε όλα τα μέσα χρηματοδότησης να ενταχθούν μέσα σε ένα συνεκτικό πλαίσιο χρηματοδότησης. Τέλος. Πάμε στους στόχους. Υπάρχουν ήδη δεσμευτικοί στόχοι α, για τις μεταφορές 10% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και 10% για τα ποιοτικά οχήματα. Με τους στόχους ε, κινούμαστε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και μετράμε και τα Προσμετράμε και τα αποτελέσματα. Αλλά αυτό δεν προδικάζει όμως τις ε, πολιτικές λύσεις. Η Κομισιόν σημειώνει με ενδιαφέρον ότι ο σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να ενταχθεί στη Λευκή Βίβλο της Κομισιόν αυτή η έκθεση. Η τελευταία μου δέσμευση για σήμερα είναι ότι θα αναλύσουμε την έκθεση και τις 376 τροπολογίες και Θα λάβουμε υπόψη όλες τις προτάσεις και τα σχολιά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γέγκε. Και ξανά ο εισηγητής μας για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ για όλες ε, τις ε, συνεισφορές. Νομίζω πως προκύπτει από τις συζητήσεις πως καλά κάναμε να αφιερώσουμε χρόνο και με τους συναδέλφους των ομάδων και με την Κομισιόν για να οριμάσουν κάποια πράγματα. Για μένα οι μεταφορές είναι το μέλλον και αυτό το οποίο είπε η συνάδελφος ισχύει πράγματι πρέπει να στραφούν προς το μέλλον οι μεταφορές και βεβαίως ε, ξέρουν οι συνάδελφοι πως ακριβώς αυτά τα θέματα που συζητάμε εδώ πέρα θα παραμείνουν στην Επιτροπή Μεταφορών. Δεν νομίζω πως χάσαμε ως ε, ε, Επιτροπή εμείς, αλλά η Κομισιόν μοίρασε έτσι τις αρμοδιότητες της, ε, έτσι ώστε θα πρέπει να αποκατασταθεί η συνοχή όσον αφορά την αντιμετώπιση των ε, μεταφορών. Για τα λεφτά. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Αυτά είναι από τους τομείς, οι μεταφορές δηλαδή, που θα ε, προσφέρουν χρήματα στα κράτη-μέλη. Είτε λέγονται τέλη, είτε λέγονται φόροι, είτε όπως αλλιώς λέγονται. Οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε σκέψη για να δούμε πώς θα γίνει αυτό με κάθε σεβασμό για την επικουρικότητα κτλ. κτλ. Ε, τι σημαίνει επικουρικότητα. Πρώτον, όταν δεν βρίσκουμε λύση, λέμε τα αφήνουμε στην επικουρικότητα ή όταν αναστατώνονται οι χώρες. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε και Πρέπει να ξέρουμε πώς υπάρχουν νέες δυνατότητες να βρουν λεφτά στις μεταφορές. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τίποτα. Υπάρχουν τα τέλη, η εξωτερικοποίηση του κόστους είναι κάτι το ενδιαφέρον και αντιλαμβάνομαι πως κάθε υπουργό Οικονομικών θα πει πως «Ε, δεν θα μου πούν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη τι θα κάνω εγώ με τα λεφτά μου, αλλά εάν χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μας ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα του προπολογισμού για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό ταμείο, τότε θα γίνει πιο ενδιαφέρουσα η συζήτηση και νομίζω πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό επιπλέον. Πράγματι δεν είναι ότι θα εφεύρουμε ξαφνικά ένα νέο φόρο. Έχουμε αρκετά μέση ήδη, αλλά πρέπει νομίζω να μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα πως οι διασυνοριακές ε, πρωτοβουλίες πρέπει να δουν το τι γίνεται και με τις υποδομές. Αν δούμε το τι έχει γίνει ε, στα τελευταία 25 χρόνια, τα τελευταία, τα τελευταία 25 χρόνια, είναι παράλογο. Π.χ στο Ταμείο Συνοχής προβλέπεται ένα ποστό για τις μεταφορές. Πρέπει να το δούμε ε, συνολικά. Επίσης, μιλήσατε για το 2009 τα 70 εκατομμύρια, 7 δισεκατομμύρια το 2010, πράγματα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να αποτελέσουν το αρχικό κεφάλαιο για συγκεκριμένα έργα, γιατί ξέρουμε ξεκάθαρα το τι λείπει. Πρώτα απ' όλα εγγυήσει μπορεί να τι σώσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και δεύτερον δεν μπορούν να γίνονται τα πάντα με χρέη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε, Μαργκερίτ, ένα ταμείο, ένα ταμείο το οποίο δεν θα χρησιμοποιήσει μόνο στην πρώτη φάση της οικοδόμηση Και τέλος εδώ πέρα να δούμε και το ιδιωτικό κεφάλαιο. Μιλάμε εδώ πέρα για ΣΔΙΤ, ε, συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Απλώς είναι ο κανόνας. Πρέπει να υπάρχει μία ελάχιστη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και κερδοφορία. Αλλιώς δεν θα έρθει ο ιδιώτης. Τώρα για την αποτελεσματική συντροπικότητα αυτή κατά την άποψή μου νομίζω δεν θέλω εγώ τώρα να δημιουργήσω νέο δόγμα, αλλά θεωρώ πως θα γίνει αναγκαστικά ένα νέο μέσο αλλαγής των μεταφορών και χρειαζόμαστε Πραγματικά και την συμπληρωματικότητα και την αμοιβαία συμπλήρωση των διαφόρων ε, μέσων μεταφοράς και χαίρομαι και για την τελευταία πρόταση της ε, Κομισιόν ε, μόλις άκουσα δηλαδή πως η Κομισιόν θα λάβει υπόψη όλες μας προτάσεις με αυτό είναι φανταστικό και αναμένω την επόμενη φάση τουλάχιστον τόσα Σαββατοκύριακα δεν εργαστήκαμε άδικα ευχαριστώ uh, Σας ευχαριστούμε κύριε Γκρός Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να περάσουμε τον Ιούνιο στην ψηφοφορία της έκθεσής σας και τον Ιούλιο στην Ολομέλεια. Εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα το απόγευμα. Μην ξεχνάτε το αυριανό μας ραντεβού στις 9 ακριβώς το πρωί με τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Παρακαλώ να τις έχετε μαζί σας. Ραντεβού λοιπόν αύριο λύεται τη συνεδρίαση για σήμερα.